Okay, colleghi, possiamo iniziare? Λοιπόν, συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. όσον αφορά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης ε, μετά από έτοιμα του κυρίου Χερντός ε, το σημείο υπαριθμών 5 της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση της έκθεσης πρωτοβουλίας που αφορά στις προοπτικές ε, και τις προκλήσεις της, του τομέα των εγωπορβάτων στην Ευρώπη αναβάλλεται. Και έτσι η ψηφορία θα λάβει η χώρα στις 23 Ιανουαρίου του 2018. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να λάβετε επίση υπόψη σα το γεγονός ότι το σημείο υπαριθμών 11 της μερίσιας διάταξης ε, που προβλέπει την παράταση των δικαιωμάτων των καλλιεργητών ε, ε, φυτών και το 12 που αφορά στην απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα θέματα αυτά αντιστρέφονται δηλαδή τα θέματα θα εξεταστούν σήμερα το απόγευμα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, σχετικά με αυτές τις ε, τροποποίησεις, θεωρούμε ότι εγκρίνεται η τροποποιημένη μερίσια διάταξη. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω διαδικτύου και επίσης να σας πω ότι η διερμηνία υπάρχει σε 20 γλώσσες, εκτός από τα τσεχικά, τα μαλτέζικα, τα σλοβάκικα και τα ε, κέλτικα. Λοιπόν, συνάδελφοι, Ξεκινάμε με, τις, ε, με την ψηφοφορία. Εν τω μεταξύ, ας ξεκινήσουμε με το σημείο υπαριθμών 3, τον κανονισμό Omnibus. Και θέλω να επενθυμίσω σε όλους σας ότι είναι ένας ε, κανονισμός ε, αυτόνομος Λοιπόν, θα ψηφίσουμε για τη συμφωνία της 12 Οκτωβρίου σχετικά με την ε, ψηφοφορία ε, Omnibus. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τα αποτελέσματα έχουν, ε, ήδη έχουν παρουσιαστεί από τον συνάδελφο κύριο από εμένα και συζητήθηκαν στην Επιτροπή Γεωργίας στις 6 Νοεμβρίου. Τώρα, η ψηφοφορία θα είναι ένα απλό ναι ή όχι όσον αφορά τα, τη δέσμη μέτρων. Ε, συνάδελφοι, ε, φαντάζομαι έχετε πάρει ένα κείμενο που αφορά ε, τις σημαντικές τροπολογίες που έλαβαν χώρα για τέσσερις, ε, βασικές, τέσσερις βασικούς κανονισμούς της κοινή πολιτικής γεωργίας. Όλα αυτά έχουν καταστήσει την αρχική πρόταση της Επιτροπής, πολύ πιο φιλόδοξη από ό,τι στάθηκε από τον Επίτροπο. Νομίζω ότι τώρα πραγματικά μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική ε, τροποποίηση μεσοπρόθεσμη τη κοινή ε, πολιτική γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω ότι μετά από την απόφαση που ελήφθη στι 16 Νοεμβρίου από τη διάσκεψη των Προέδρων, ε, μία τροποποίηση που αφορά το να αφαιρεθεί αυτή η τροπολογία από το υπόλοιπο πακέτο, η Επιτροπή Γεωργίας έγινε η επί της αρμόδια επιτροπή για το πρώτο κομμάτι του κανονισμού. Ως εκ τούτου αυτό θα αντιμετωπιστεί ως ένας αυτόνομος κανονισμός. Και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον γιατί εκτός από το περιεχόμενο και από πλευράς διαδικαστικής αυτή η Επιτροπή ε, χάραξε ένα, μια καινοτόμα πορεία, αλλά κυρίως μια πορεία που μας επιτρέπει να θέσουμε σε ισχύ αυτή τη δέσμη μέτρων από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Πριν λοιπόν από την ψηφοφορία θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Άλμπερντες. Παρακαλώ Αλμπερντ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Πάολο, αγαπητέ Πάολο, θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους ε, όσοι συνέβαλαν ε, στις εργασίες μας. Τρεις τριμερείς διαλόγους είχαμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεκάστρο και τον Μίχαλ Νταντό αλλά και όλους τους άλλους σκιώδεις συγητές, να ευχαριστήσω συνεργάτες να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο και επίση και όλους εκείνους ε, ε, που συνεργάστηκαν στην Επιτροπή. Γιατί ε, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να έχουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις και θέλω να σας πω ότι η συνεργασία ήταν ιδιαίτερα αγαστή και ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Υπάρχει τώρα πλέον αυτή η διαδικασία ε, και ευχαριστώ και την κυρία Κρέσλε που συμφώνησε όλα αυτά να γίνουν ξεχωριστά. Την τελευταία στιγμή γίναν όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγιναν και ε, το όλο θέμα μπορεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου. Κοίτα, δεν μπορώ να κατεβάσω την ψηφοφορία, πίστευτο. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, ως εκ τούτου ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε ψηφοφορία. «39 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, εγκρίναμε τον κανονισμό για τη μεταρρύθμιση της κοινή πολιτικής γεωργίας. Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, προχωράμε στο σημείο υπαριθμών 4 της ημερήσιας διάταξης. Η βιολογική παραγωγή ε, προχωράμε λοιπόν στην ψηφοφορία που αφορά στον κανισμό σχετικά με την ε, βιολογική παραγωγή και την ετικετοθεσία οργανικών προϊόντων. Όπως ξέρετε, στις 20 Νοεμβρίου η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε την ε, συμφωνία που επιτέχθηκε στις, ε, στον τριμερή διάλογο 18, Ιουλίου, 18 Ιουνίου 2017. Και πριν ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, θα ψηφίσουμε εδώ για το ενοποιημένο κείμενο. Μία και μόνο ψηφοφορία θα έχουμε, όπως κάναμε και με την ψηφορία για τον κανονισμό Omnibus. Αν ο Μάρτιν θέλει να λάβει το λόγο, παρακαλώ Μάρτιν, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Πράγματι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορούμε να πούμε ότι το Συμβούλιο συμφώνησε. Ε, έχουμε μια νέα πρόταση, την πήραμε Δευτέρα, 279 σελίδες. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους σκιώδης ηγητές. Ήταν μια πολύ καλή συνεργασία εμείς ε, τις δικές μας προτάσεις μπορέσαμε να τις ε, περάσουμε. Θέλω λοιπόν να ελπίζω ότι το θέμα αυτό θα ολοκληρωθεί με μεγάλη ε, ψηφοφορία, με μεγάλη πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ για την αγαστή συνεργασία και ελπίζω να υπερψηφιστεί η πρότασή μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Μάρτιν. Προχωράμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία και εδώ μία μόνο ψηφοφορία, ναι ή όχι. Πρόταση ηλεκτρονικής ε, ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε παρακαλώ για τη δέσμη μέτρων. Chiaro chiusa la Approvato. Λοιπόν, εγκρίθηκε 29 υπέρ, 11 κατά, 4 ε, αποχές και εγκρίθηκε ε, άρα <clears throat> το όλο θέμα θα πάει στην Ολομέλεια. Ναι. Α, το 5 είπα να βάλω, την πάμε E λοιπόν, συνάδελφοι, προχωράμε με τη συζήτηση για το σημείο υπερθμών 6 ε, το σημείο 6, η τρέχουσα κατάσταση και οι μελλοντικέ προοπτικές για τον ε, τομέα των εγωπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτρια, η Εστεχεράντς Χεράνς Γκαρσία, <clears throat> παρακαλώ, θα λάβετε το λόγο, γιατί εδώ πρόκειται για ένα από τους πιο ευαίσθητους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και θα αντιμετωπίσει κυρίως ε, τις επιπτώσεις από το Brexit. Η συγγήτριά μας, η κυρία Γκαρσία, θα μας παρουσιάσει σήμερα το σχέδιο της έκθεσης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία Χεράντς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι τη φασαρία που γίνεται, γιατί μετά από δύο χρόνια συζητήσεις για τα βιολογικά προϊόντα, επιτέλους ε, εγκρίναμε τη σχετική πρόταση, οπότε είναι φυσικό να υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Εμείς περνάμε τώρα στα εγωπρόβατα, ένα πολύ σημαντικό κλάδο παραγωγής ε, για τις αγροτικές ζώνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα από τους πιο έφθραυστους ε, και ευάλωτους κτηνοτροφικούς κλάδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επίπεδο εγκατάλειψης, η γύρες των επαγγελματιών, η μείωση της ε, κτηνοτροφικής παραγωγής και η εξάρτηση των κτηνοτρόφων αυτών από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ καθιστούν τον κλάδο πολύ ευάλωτο και θα πρέπει να τον φροντίσουμε με ιδιαίτερη στοργή. Ήδη είχαμε κάνει ε, μια προκαταρκτική συζήτηση για αυτή την έκθεση πρωτοβουλία και νομίζω ότι συμφωνούν οι συνάδελφοι και πιστεύω ότι θα έχουμε αγαστή και πολύ στενή συνεργασία για το έγγραφο που θα σας παρουσιάσω. Όπως ξέρετε, το σύνολο του κλάδου της εγωπροβατοτροφίας ε, είναι σημαντικό. Βέβαια, ο μεγαλύτερο παραγωγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγωπρόβιου κρέατο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε το Brexit θα έχει σημαντικέ επιπτώσει στι εμπορικέ ροέ. Επιπλέον, έχουμε τι περικοπέ στον προπολογισμό. που είναι αναμενόμενες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά το Brexit. Το Brexit λοιπόν θα επηρεάσει διπλά τον κλάδο της εγωπροβατοτροφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενός το Ηνωμένο Βασίλειο είναι βασικός παραγωγός εγωπρόβιου κρέατος και αφετέρου με την αποχώρησή του θα, θα συρρυκνωθεί ο προϋπολογισμός. Άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το επίπεδο αυτάρκειας. Δεν παράγουμε αρκετό εγωπρόβιο κρέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψουμε τις ανάγκες καταναλωτικές μας. Οπότε ε, και επιπλέον οι ανταγωνιστές μας, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, μας στέλνουν ε, τα ε, εμπορεύματά τους σε τις περιόδους της εχμής, δηλαδή Χριστούγεννα ή Μεγάλη Εβδομάδα ενώπιση του Πάσχα, που είναι και η περίοδη της μεγαλύτερης κατανάλωσης. Επίσης, έχουμε προβλήματα με τους θηρευτές, λύκους, αρκούδες. Το αντιμετωπίσαμε το θέμα αυτό και σε άλλη γνωμοδότηση, αλλά ακόμη δεν έχει ε, λυθεί το πρόβλημα των θηρευτών που αποδεκατίζουν τα πίμνια. ήδη ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησε ένα φόρουμ για το γοπρόβιο κρέας το 2015 που ήταν πολύ σημαντική πλατφόρμα συζητήσεων για τον κλάδο. Και μάλιστα εμεί σηκώνουμε το γάντι που μας στέλνει το φόρουμ αυτό για το γοπρόβιο κρέας και με την έκθεση του θέλουμε οι κτηνοτρόφοι μας να βελτιώσουν την ε, διαπραγματευτική τους θέση στην τροφική αλυσίδα, να διαφυλάξουμε αυτό το κλάδο και αν γίνεται να τον ενισχύσουμε κιόλα. να το δώσουμε μια μελλοντική προοπτική και γι' αυτό θα πρέπει να το στηρίξουμε σε όλες τις φάσεις, στην ε, επένδυση, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, να στηρίξουμε τους νέους κτηνοτρόφους που θέλουν ε, να, να ξεκινήσουν με τα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου και με τις ειδικέ ενισχύσεις στην εγωπροβατοτροφία και επίσης να δώσουμε κίνητρα για την ανανέωση των γενεών και στην κτηνοτροφία. Επίσης, να σκεφτούμε και ίσως και μία ειδική ενίσχυση. Είναι πολύ διάζων αυτός ο κλάδος, γιατί πραγματοποιεί μία περιβαλλοντική υπηρεσία άνευ προηγουμένου για τον κλάδο. Γιατί ειδικά η εγωτροφία έχει σημαντική περιβαλλοντική αξία και μάλιστα αναντικατάσταση, αναντικατάστατη. Και δυστυχώς με τη συρρήκνωση των ποινίων χάνουμε αυτή την περιβαλλοντική υπηρεσία που γίνεται στους βοσκοτόπους ιδιαίτερα ε, όταν ε, βοσκούν έγες. Γι' αυτό ε, μιλούμε για περιβαλλοντικά μέτρα, μα η εγωτροφία τα πραγματοποιεί. Αν λοιπόν δεν είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν ε, αντιμετωπίσουμε με στοργή τον κλάδο, θα χάσουμε, θα χάσουμε και την θετική περιβαλλοντική επίπτωση. Θα μπορούσα να σας απαριθμίσω και τα υπόλοιπα μέτρα που προτείνω, αλλά προτιμώ να ακούσω τις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις και είμαι στη διάθεσή σας για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση. Έχουν ζητήσει το λόγο διάφοροι συνάδελφοι. Ο Ερικ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ και με την ανάλυση του προβλήματος που κάνει και με τις λύσεις που προτείνει. Πράγματι πρέπει να βρεθεί μια νέα ισορροπία στις ενισχύσει που δίνονται στον τομέα της πρόβατοτροφίας γιατί υπάρχουν περιοχές με, ε, ε, ε, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και θα πρέπει να τις βοηθήσουμε ιδιαίτερα, να βοηθήσουμε ιδιαίτερα επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, σε αυτές τις περιοχές. γιατί αυτός ο τομέας βοηθάει την καταπολέμηση της ανεργίας σε αυτές τις περιοχές και όπως είπατε και το περιβάλλον. Είναι ένας... Είναι και οι δύο τομείς πολύ σημαντικοί. Και Πιστεύω ότι επίση το ζήτημα τη γαλακτοκομία πρέπει να το αναδείξουμε, γιατί γενικά μιλώντα για την εγωπροβατοτροφία ε, έχουμε τον τομέα του γάλακτο και τον τομέα του κρέατο. Πρέπει να νομίζω να αναδείξουμε και το ζήτημα του γάλακτο. Πρόκειται για έναν τομέα της οικονομίας που έχει μια σημαντική προστιθέμενη αξία. Το βλέπουμε αυτό στις περιοχές της Γαλλίας που, όπου διαραστηριοποιείται ο κόσμος στον τομέα αυτόν. Πρόκειται για τομείς της οικονομίας ευαίσθητους και επομένως θα πρέπει να φροντίσουμε να τους στηρίξουμε τα επόμενα χρόνια. Και όπως είπατε πράγματι υπάρχει και το ζήτημα των θηρευτών, ιδιαίτερα των λύκων που δημιουργεί προβλήματα για την ανάπτυξη του κλάδου αυτού. Ίσως θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια ομάδα προβληματισμού, μια ομάδα για τους λύκους συγκεκριμένα, για να δει πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ε, ε, ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο εμποδίζει την σωστή ανάπτυξη του κλάδου αυτού και το αντιμετωπίζουμε και σε πολλές χώρες, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Ιδιαίτερα στο, στην περιοχή της Μεσογείου. Το νερό είναι διαχείριση των υδάτινων πόρων, λοιπόν, ειδικά στη Μεσόγειο, ειδικά στο Νότο, είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Εράνς Καρσία γιατί έχει ήδη κάνει σημαντική προεργασία και βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο της επεξεργασίας της ε, έκθεσής της. Συμφωνώ με τον κύριο Αντριέ και με την εισηγήτρια ως προς τη φιλοσοφία που αναπτύσσει και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε από κοινού να συντάξουμε τροπολογίες για να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε το κείμενο. Πάντως το θέμα του γάλακτος ε, έχει κέριο ρόλο φυσικά στα πρόβατα αλλά ακόμη περισσότερο στα ερήφια, στην εγωτροφία, γιατί 90% των, ε, της θηροκομικής παραγωγής για πρόβιο και κατσική κρέας είναι από γίνεται από τρεις χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, γεωγραφικές ενδείξεις για το κρέας ε, του αμνού, που δεν ε, τις προασπίζουμε στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουμε. Και θα ήταν πολύ σημαντικό να ληφθεί και αυτό υπόψη. Επίσης, θα πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα όλο το θέμα της γαλακτοκομικής μας παραγωγής από πρόβατα. Επίσης, τονίστηκε πολύ σωστά ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Γιατί λοιπόν να μην προτείνουμε μία πρακτική ιδιαίτερα για την εγωτροφία που θα συνδέεται περισσότερο με τα λιβάδια, με, τα... με τους βοσκοτόπους γιατί έχει πάρει τον κατήφορο δυστυχώς ε, η εγωτροφία και γίνεται εκτός του, των στάβλων ε, α, ή μάλλον ε, με, μέσα στους στάβλους χωρίς να έχουν επαφή με, τη, με τα βοσκοτόπια. Θα πρέπει να έχουμε πιο εκτατική εγωτροφία, να βοσκούν στα λιβάδια οι έγες. Και όσο σε ό,τι αφορά τους θηρευτές και εκεί θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη πυγμή, γιατί στην Ισπανία το 2016 είχαμε 4.600 επιθέσεις από Δυστυχώς δεν έχει μειωθεί αυτός ο αριθμός. Ίσως θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι στο ρόλο της συνθήκης της Βέρνης και ε, να το συνδυάσουμε με την οδηγία μας για τα ενδιατήματα και να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι και σαφείς. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα κινηθούμε και στις τροπολογίες σε, στην ίδια γραμμή πλεύση με την εισηγήτρια, η έκθεση της οποίας βαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρντος. Δεν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική εκθέση που έχει προετοιμάσει και να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα που έχει συμπεριλάβει και τις δικές μου προτάσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τη στήριξη των παραγωγών. και των κτηνοτρόφων. Κατά την άποψή μου, η στήριξη των παραγωγών θα πρέπει να απευθύνεται σε, διαφορετικές, σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες ε, κτηνοτρόφων θα μπορούσε να είναι ένα εφάπαξ ποσό, ένα καταποκοπήν ποσό για τους μικρούς παραγωγούς, τις μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω από 15 ζώα και ε, μια πιο προοδευτική στήριξη των μεγαλύτερων ε, κτηνοτροφικών μονάδων. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα ε, μέσα στήριξης της γαλακτοκομικής των παραγωγών, όλα αυτά τα μέσα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για, την, α, για τους παραγωγούς γάλακτος από ερήφια. Ε, επίσης πρέπει να συμπεριληφθούν τα ε, ζώα αυτά και στις, στα μέσα που έχουμε για την στήριξη των μέτρων ε, υπέρ της ευζοίας των ζώων. Ο, τα, τα, τα, χρήματα που είναι διαθέσιμα στην ΚΑΠ για αυτού του τύπου τα μέτρα ε, μειώνονται διαρκώς και πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί <clears throat> έτσι ώστε να ε, εντοπιστούν που είναι πραγματικές ανάγκες. Πρέπει να δούμε επίσης την εκπαίδευση ε, επιμενικών σκύλων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κοινοτρόφους για να προστατεύσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς θα φροντίσουμε για την ισότητα των δύο φύλων, πώς θα φροντίσουμε περισσότερες γυναίκες να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτόν. Είμαστε πια στον 21ο αιώνα και οι γυναίκε και οι άνδρε μπορούν εξίσου να ασχοληθούν με τον κτηνοτροφικό τομέα. Αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ζαν Πολ Ντενανό έχει το λόγο. Και μετά η κυρία Γκυλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω το έργο της συγκεκριτήρια τη κυρία Εράς Γκαρσία και να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο κυρίως θέματα. Το πρώτο αφορά τους γενετικούς σπόρους που είναι σημαντικοί για την ε, ποιοτική παραγωγικότητα και την ε, διατήρηση σημαντικών ε, παραδοσιακών φυλών ζώων. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να το λάβουμε υπόψη στο μηχανισμό επιλογής το θέμα της προσαρμογής των ζώων και το γονότυπό τους. Επίσης το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων, πολύ σημαντικό και βέβαια η εγωπροβατοτροφία μάλλον είναι υπέρ της καλής μεταχείρισης, προσφέρεται για καλή μεταχείριση των ζώων. Επίσης, ε, το συγχρονισμό ε, σε περίπτωση ε, εγγύων ζώων που εισάγονται από την Ουρουάη και άλλες χώρες. Θα πρέπει να μην διαταράσει αυτό τον κύκλο των ντόπιων ζών. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για, τους, για τον κλάδο της εγωπροφωτοτροφίας. Επίσης το θέμα των βοσκοτόπων. Θα πρέπει κάποιες ζώνες ε, να τις διαφυλάξουμε για τη χορτονομία, για, να επιτρέψουμε τέτοια εκτατική εγωπροβατοτροφία στο φυσικό περιβάλλον που είναι οι βοσκότοποι. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγιλέρα. Κλάρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τη Εστέρ Εράνς Γκαρσία για την καλή της έκθεση. Η Ισπανία είναι μια χώρα με σημαντική εγωπροβατοτροφία και δεν με εκπλήσει που είναι πραγματικά άρτη η έκθεση της κυρίας Ερά Γκαρσία γιατί ε, γνωρίζει τον κλάδο, είναι εξοικειωμένη με τα προβλήματά του και μπορεί να θεωρείται ίσως σημασία σε αυτού του είδους η κτηνοτροφία, αλλά η σημασία της για τους ε, τοπικούς πληθυσμούς, αλλά και για το περιβάλλον είναι πολύ σημαντική. Επαναλαμβάνω, η έκθεση, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ καλή. Μερικά θέματα που θα καταθέσω εδώ και θα τα περιλάβω και σε τροπολογίες είναι τα εξή. Κατά τη γνώμη μου, σε μια έκθεση για την εγωπρόβατοτροφία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εκτατική κτηνοτροφία. Δηλαδή το είδος της κτηνοτροφίας που γίνεται στους αγρούς, στα λιβάδια, σε συγκεκριμένα οικοσυστήματα που συνάδει με την διαφύλαξη αυτών των οικοσυστημάτων. Πρόκειται για μια κτηνοτροφία ιδιαίτερα στην περίπτωση των εγωπροβάτων που καλό θα ήταν να, λάβει προτεραιότητα και στις ενισχύσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εγώ πιστεύω στην εκτατική κτηνοτροφία, γιατί θεωρώ ότι το περιβαλλοντικό της όφελος είναι υψηλό και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα και με οικονομική στήριξη σε αυτή την εκτατική κτηνοτροφία, ιδιαίτερα την εκτατική εγωπροβατοτροφία. Επίσης, να αναδείξουμε και να αναβαθίσουμε αυτά τα προϊόντα για να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους. Για παράδειγμα, το μαλλί, το δέρμα, να αξιοποιήσουμε το μαλλί και το δέρμα που είναι υποπροϊόντα αυτής της κτηνοτροφίας. Έτσι αναβαθμίζουμε και αναδεικνύουμε τα ωφέλη αυτού του είδους της κτηνοτροφίας που αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες και αντικσότητες και εξαφανίζεται σταδιακά από τα τοπία μας. Επίσης, η κατάρτιση των ποιμένων είναι πολύ σημαντικό. Ε, φαίνεται κάτι εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί ελάχιστοι αρχίζουν και ασχολούνται με τέτοιου είδους ε, κτηνοτροφία. Και όταν ε, αρχίζουν την εγωπροβατοτροφία κάποιοι νέοι, δεν ξέρουν πώς θα το χειριστούν. Στην Ανδαλουσία έχουμε σχολή ποιμένων, σχολή βοσκών, και είναι σημαντικό να καταρτίζουμε τους νέους για τις δραστηριότητες και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια. Ε, δεν είναι αρκετά γενικευμένη η κατάρτιση των ποιημένων, γιατί έχει ειδικά χαρακτηριστικά και ειδικέ ανάγκε, χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση. Θα πρέπει να καταρτίζονται λοιπόν σωστά οι βοσκοί. Επίσης, ε, ε, για την περικοπή που θα γίνει τη δημοσιονομική. Γνωρίζω, Εστέρ, ότι όλοι θα δώσουμε μάχη μέχρι τελική ρανίδο για να μην περικοπεί ο γεωργικό προπολογισμό ούτε, ούτε κατά ένα ευρώ. Και δεν μου αρέσει να το συζητάμε ήδη και να ξεκινάμε από αυτό το τεκμήριο ότι θα έχουμε de facto συρρήκνωση ή περικοπή του γεωργικού προπολογισμού. Στο παρελθόν ασχοληθήκαμε το θέμα των θηρευτών και ιδιαίτερα των επιθέσεων λύκων σε μια γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, που ψηφίσαμε κατά γιατί τέτοιου είδους ε, επιθέσεις από θηρευτές επηρεάζουν ιδιαίτερα τέτοιου είδους κτηνοτροφία. Ο Μάρκ Ταραμπέλα και μετά η κυρία Σένρα. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που επένασαν την εισηγητριά μας, την κυρία Ράς Καρσία. Εγώ θα σταθώ σε δύο σημεία. Το πρώτο που αναφέρεται στις παραγράφους 9, 10 και 11 και στην αιτιολογική έκθεση αφορά τις συνέπειες του Brexit. Καταρχήν από χώρε όπως η Αργεντινή, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδάς, Ουρουγουάη που τα μεταφέρουν το προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμή μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου πώς θα γίνει κατανομή, ανακατανομή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά εδώ έχουμε και ευκαιρίες που θα πρέπει να δράξουμε και ίσως αυτό το το θετικό ε, αποτέλεσμα που θα έχει το Brexit να το αξιοποιήσουμε και εμείς. Επίσης, ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο όταν εισήλθε το 1973 διεκδίκησε κάποια πλεονεκτήματα για τις παλιές χώρες της κοινοπολιτείας. Από τη στιγμή όμως που θα αποχωρήσει και αποφάσισε να αποχωρήσει με πλειοψηφία του πληθυσμού το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα που είχαμε δώσει στις χώρες της κοινοπολιτείας. Ε, γιατί να μην ε, αυξήσουμε τις, ε, την παραγωγή μας στις υπόλοιπες 27 χώρες, στην Ιρλανδία που θα πληγεί ιδιαίτερα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειου, αλλά και στις υπόλοιπες. Προσοχή λοιπόν να μην ενδώσουμε ή να μην μυρολατρούμε σε ό,τι αφορά τις συνέπειες του Brexit και να μην σταθούμε μόνο στα αρνητικά χαρακτηριστικά. Επίσης μπορούμε να ενθαρρύνουμε την αγαπροβατοτροφία, ιδιαίτερα στις μειονεκτικές ζώνες που δεν είναι δυνατά άλλα είδη γεωργίας εκτινοτροφίας, Ζητώντα συνδεδεμένε ενισχύσει για, τη, για την εκοπροβοτοτροφία στην επόμενη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ και επίση να έχουμε μια αιρεσιμότητα που θα συνδέεται με το έδαφο. για να μην ενθαρρύνουμε βιομηχανική κτηνοτροφία που θα είναι αντιπαραγωγική και δυσμενή για το περιβάλλον. Μπορεί να έχουμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια, δηλαδή και να αυξήσουμε την παραγωγή εγωπρόβιου κρέατος στις υπόλοιπες 27 χώρες, με αύξηση της εκτατικής κτηνοτροφίας όμως, που θα σέβεται και την περιβαλλοντική αιρεσιμότητα και κυρίως θα ενισχύει τις ε, πλέον μειονεκτούσες αγροτικές περιοχές που πολύ συχνά είναι τα θύματα της εγκατάλειψης του πληθυσμού και της απερίμωσης. Η κυρία Σένερα και μετά ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ. Πρώτα κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Εστέρ για την προσπάθειά της, για το έργο της. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό σημείο η έκθεσή της και πιστεύω, όπως θα πω και στις τροπολογίες μου, ότι καλό θα είναι να σταθούμε περισσότερο στο, στο θέμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της βιοπικιλότητας που προσφέρουν η κλάδη της ε, κτηνοτροφίας ε, εγώ και προβάτων. Και σε ό,τι φορά τη Γαλλικία, ε, πολύ σημαντικό θα ήταν να στηρίξουμε την εγώ προβατοτροφία, γιατί είμαστε θύματα συχνών δασικών πυρκαγιών και το θέμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής φροντίδας ή της στήριξης του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει να στηρίξουμε τις αυτόχθονες φυλές ζώων που έχουν πολύ μεγαλύτερες ικανότητες για να προσαρμόζονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Επίσης, να στηρίξουμε τα γεωργικά εισοδήματα των απασχολουμένων στον κλάδο αυτό της κτηνοτροφίας. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό σε δύο επίπεδα. Να έχουμε μηχανισμούς για τη βελτίωση των τιμών ε, στον παραγωγό και επιπλέον να αναλύσουμε ε, τις δυσκολίες ώστε να δώσουμε έμφαση στις άμεσες πωλήσει και στην, ε, ε, στο εμπόριο σε πολύ στενό κύκλο, σε πολύ μικρές αποστάσεις. Επίσης να αναλύσουμε τον αντίκτυπο των θηρευτών στα πίμνια. Και εκεί που υπάρχουν βοήθειες, ενισχύσεις στον κλάδο είναι καταρχήν ελάχιστες και επίσης ε, καταβάλλονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν αυτά που είπα και οι συνάδελφοι και τις υπόλοιπες δυσκολίες. Ε, συμφωνώ και σταματώ εδώ. Κύριος Ντόρφμαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Έστερ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και πράγματι είναι αλήθεια ότι η εκτατική εγωπροβατοτροφία, κυρίως στις ορεινές περιοχές, είναι μια σημαντική πηγή εισοδήματος. Γι' αυτό λοιπόν πολύ σωστά συζητάμε για το θέμα αυτό για άλλη μια φορά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Έστερ θίγει και το θέμα των θηρευτών, κυρίως των λύκων. Εγώ θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια πολύ σημαντική ψηφοφορία στην Ολομέλεια ε, και εκεί νομίζω επιτύχαμε και μια ρήξη με το παρελθόν διότι επιτύχαμε δια κομματική συμφωνία συμφώνησαν δηλαδή όλε τι πολιτικέ ομάδε και ω εκ τούτου οφείλουμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να κατατεθούν συγκεκριμένε προτάσει. Γιατί μέχρι τώρα μα καθυστερούν και μα λένε ότι υποτίθεται υπάρχουν κάποια καλά μοντέλα συμβίωση. Εγώ όμω δεν τα έχω δει. Πού υπάρχουν αυτά. Εγώ δεν τι βρίσκω αυτέ τι περιοχέ όπου υποτίθεται ότι υπάρχει μια ικανοποιητική συμβίωση ανάμεσα σε μικρά ζώα και λύκους. Ε, άρα πρέπει να σκίσουμε πίεση και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εγωπροβατοτροφία σε περιοχές με αγέλες λύκων αυτό δεν μπορεί να υπάρξει, δεν υπάρχει ε, καλή συμβίωση, προκύπτουν δυσκολίες, η συνύπαρξη δεν είναι δυνατή. Ως ε, εκ τούτου, αν συνεχίσουμε αυτή τη στάση, θα εξαφανιστεί η εγωπροβατοτροφία και δεν πρέπει αυτό να το ρισκάρουμε η ε, κυρία Μούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για αυτή την πολύ καλή έκθεση. Φύγει πολλά θέματα. Εγώ πιστεύω ότι πολύ μικρή ε, εκτροφής εγών και προβάτων με την εκτροφή ε, κάποιων ιδιαίτερων φυλών επιθυμούν να διατηρήσουν ε, τις επιχειρήσεις τους. Για μένα είναι σημαντικό στις Αλπείς ε, να υπάρχει ένας χώρος όπου να δραστηριοποιούνται μόνο εκτροφής εγών και προβάτων και να έχουμε εγγυήσει γι' αυτό. Έχω και εγώ επιφυλάξεις τις ίδιες ε, που εξέφρασε ο προλαλής σχετικά με τους λύκους και τους μεγάλους ε, θηρευτές. Ε, πρόσφατα 40 ε, πρόβατα χάσαμε. Νομίζω λοιπόν ότι ούτε τα προστατευτικά σκυλιά ούτε οι φράχτες επιφέρουν αποτέλεσμα. Σε συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να σκεφτούμε να έχουμε περιοχές χωρίς λύκους που να προστατεύονται από λύκους. Ε, τα προγράμματα ε, στα χαρτιά δεν λύνουν τα προβλήματα και οι υβριδιακές καταστάσεις ε, επιτείνουν το πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτήν την έκθεση έχουμε πολύ καλά σημεία τα οποία ε, προστατεύουν τις έγες και τα πρόβατα κυρίως στο δεύτερο πυλώνα όπου λέμε ότι οφείλουμε να προβλέψουμε μεγαλύτερες ενισχύσεις για τους ε, εγωπροβατοτρόφους. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η κλάδη της εκτροφής εγών και προβάτων και μάλιστα δυστυχώς ε, τους αγνοούμε ε, σε σχέση με τα βοήδη για παράδειγμα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Και ένα από τα αίτια αυτής της έλλειψης είναι το γεγονός ότι ε, προβατοτροφία γίνεται συνήθως σε αεροκατοικημένες περιοχές και απόμακρες. Αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα και στη Ρουμανία. Πολλοί εκτροφείς εγών και προβάτων εγκαταλείπουν ε, τις ε, εκμεταλλεύσεις τους εξαιτία αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν την απασχόληση στον κλάδο. Επίση, θα πρέπει να στηρίξουμε τον κλάδο και με άμεσε ενισχύσει. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την εγωπροβατοτροφία όπως και την εκτροφή βοηδών. Επίσης να δούμε το μέγεθος αυτών των άμεσων ενισχύσεων και να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι ε, οι εγωπροβατοτρόφοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τους λοιπούς κτηνοτρόφους, ιδιαίτερα τους εκτροφείς βοηδών. Ας μην ξεχνούμε ότι η ειδική αυτή κτηνοτροφία ε, γίνεται συνήθως σε απόμακρες περιοχές, ε, μειονεκτικές, με πολλές αντικσότητες. Γι' αυτό θα πρέπει να προβλέψουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα για αυτούς τους κτηνοτρόφους. Με ανησυχεί πολύ η συζήτηση που γίνεται τελευταία για τις εισαγωγές και την αύξηση των εισαγωγών τέτοιου κρέατος από τη Νέα Ζηλανδία και τις χώρες του Μερκοσούρ. Φαίνεται όμως να αγνοούμε ε, το γεγονό ότι οι χώρε αυτέ δεν επιβάλλουν του ίδιου ε, περιορισμού και τι ίδιε προδιαγραφέ ε, στου γεωργού του. Οι Ευρωπαίοι, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι υπακούν σε μια πολύ αυστηρή νομοθεσία, με πολύ ψηλά πρότυπα και προδιαγραφέ. Αυτό είναι άδικο λοιπόν για αυτού. Γιατί όταν εισάγουμε κρέα από άλλε περιοχέ του κόσμου, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί των τρίτων χωρών δεν υπάγονται στις ίδιους όρους. Οπότε η παραγωγή κρέατος γίνεται πολύ διαφορετικές συνθήκες από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπεν. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η έκθεση και έρχεται και σε, ένα, ε, σε μια σωστή χρονική στιγμή και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία μας. Πώς γνωρίζετε, πολλές χώρες στην Ευρώπη, ανάμεσα τους και η Πολωνία, έχουν αντιμετωπίσει ε, προβλήματα από την γρήπη των χείρων και έχουν στραφεί σε πολλές περιπτώσεις σε εναλλακτικές ε, επιλογές στην, στην κτηνοτροφία και αντί να, να, να παράγουν χείρους, για παράδειγμα, έχουν επιλέξει να περάσουν στα πρόβατα. Αυτό έχει συμβεί σε διάφορες χώρες, ανάμεσα σε αυτές και στη Λουθανία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας και να τον υποστηρίξουμε περισσότερο. Πριν από 50 χρόνια η τροφία είχε πολύ, μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη σημασία. Και ενώ τα τελευταία χρόνια τον έχουμε κάπως ομελήσει τον τομέα αυτόν. Και αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Το βλέπουμε παντού, το βλέπουμε και στη Λιθουανία. Όταν αυξήθηκε η κτηνοτροφία των προβάτων, ε, αρχίσαν να διαπιστώνουν ότι υπάρχουν και μεγαλύτερα προβλήματα με, τους, με τις επιθέσεις λύκων. Στο ζήτημα ιδιαίτερα των λύκων πιστεύω θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε κάποιες ε, ε, πρόοδους στην τεχνολογία. Για παράδειγμα το, τα τσιπάκια σε, στα, στα ζώα, στους, στους λύκους προκειμένου. Ίσως θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε αυτό δυνατότητα με κάποια πιλωτικά προγράμματα. Πριν από λίγες εβδομάδες διαβάσαμε στις ειδήσει ότι αγέλες λύκων επιτέθηκαν σε πρόβατα που βρίσκονταν ε, μέσα στο, στο, στο στάβλο είχαμε. Ε, και τέτοια περιστατικά. Αυτό που διαπιστώνω πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη στους κτηνοτρόφους που θέλουν να προστατευτούν από τις επιθέσεις των λύκων. Ευχαριστώ κύριο Σάκνιο. Διαπίστωσα ότι δεν αναφέρεται μία χώρα σε όλη αυτή τη συζήτηση και σε αυτή την έκθεση, η Κίνα. Και η, η, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία είναι χώρες με τις οποίες ε, η Κίνα κάνει, ε, έχει εμπορικές ε, συναλλαγές το οποίο σημαίνει ότι τα πρόβατα τα οποία δεν τα στέλνουν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία που πουλούν στην Ευρώπη τα πουλούν στην Κίνα. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία εδώ. Κάτι ακόμα είναι τα, τα γυρασμένα ζώα, τα οποία έχουν, ε, έχουν έχει αυξηθεί η αξία τους, αν συγκρίνω με το πώς είχαν τα, με τα πράγματα στο παρελθόν αναφέρθηκε, αναφέρθηκαν οι επιπτώσεις του Brexit και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στα εγωπρόβατα. Ναι, αλλά υπάρχει και το αντίστροφο επιχείρημα και οι ε, Γάλλοι παραγωγοί κρασιού θέλουν να πολλούν τα προϊόντα τους στην Αγγλία και το ίδιο ισχύει για τους Ισπανούς που θέλουν να πολλούν τα φρούτα τους. Πρέπει να βρούμε λοιπόν λύσεις που να βασίζονται στη λογική. Ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους χώρους οικολογικής εστίασης αυτές τις μορφές. Χρειάζεται να ναι, να, να, να, να αξιοποιηθούν και οι θετικές επιθέσεις που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον αυτές τις πρακτικές. Τα, το, τα συστήματα που έχουμε για την παρακολούθηση τώρα δεν λειτουργούν. Αναφέρθηκαν τα ζητήματα του περιβάλλοντος και το πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα εγωπρόβατα για το περιβάλλον. Ε, ε, προσέχοντας βέβαια να μην οδηγείται κανείς στην αποψήλωση του βοσκοτόπου. Επίσης, οι πρακτικές κτηνοτροφίας, όπου μερικές φορές είναι κλεισμένα τα εγωπρόβατα και δεν βγαίνουν ποτέ στη φύση, Θέλετε να σταματήσω κύριε Πρόεδρε γιατί μου δώσατε τρία λεπτά και θα επιμείνω να τα αξιοποιήσω και τα τρία. Όχι, να σταματήσω τώρα. Συγγνώμη. Ο κύριος Λοαζό και μετά ο κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον. Συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τον τομέα και μάλιστα είχα πει και στην ε, Κομισιόν πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος ε, που ε, συμβάλλει πολύ και στην προσθέση του περιβάλλοντος, να μην ξεχνάμε το ρόλο των λιβαδιών, έχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Επίσης, δυστυχώς, πολλοί κτηνοτρόφοι χρειάζεται να καταλήψουν τη δραστηριότητα γιατί τους πιέζουν οι τράπεζες και υφίστανται ε, ισχυρό ανταγωνισμό και πολύ σωστά ε, δακτυλοδεικνύεται τον ε, ανταγωνισμό από την Νέα δηλαδή κάτι που αποδεικνύει την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος εμποδίζει τον προστατευτισμό, ποιος ευνοεί την εγκληματική αυτή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που θα είναι ολέθρια για τον κλάδο εγωπροβάτων. Διαβάζοντας λοιπόν ε, την έκθεση διαπιστώνουμε μία μόνο λύση υπάρχει, να ζητήσουμε να σταματήσουν οι εισαγωγές ή να επιβάλλουμε φορολογία που θα ευνοεί την ευρωπαϊκή παραγωγή και φυσικά να διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Επιθυμεί όμως κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ αμφιβάλλω. Οπότε αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον πια η έκθεση. Ευχαριστώ κύριο Φλάναγκαν. Uh, Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την έκθεση. Έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και ιδιαίτερα για το τελευταίο ζήτημα που συζητάμε, το Omnibus, όπου τίθεται το θέμα των ποιων περιοχών θα είναι επιλέξιμες, νομίζω ότι είναι και αυτό ένα ζήτημα που ιδιαίτερα ενδιαφέρει τους κτηνοτρόφους, γιατί χρειάζονται μια υποστήριξη αυτή οι κτηνοτρόφοι. Έχουμε τα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα υποστήριξης όσο είναι πάρα πολύ περίπλοκα ε, και φαίνεται ότι το πρόβλημα επηρεάζει τους κτηνοτρόφους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα προβλήματά τους είναι ότι δεν έχουν καλή εκπροσώπηση στις διάφορες διαπραγματεύσεις και αυτό πρέπει να αλλάξει στο μέλλον, ελπίζω. Ε, βασίζονται μονάχα στον πυλώνα 2 της ΚΑΠ και θα, θα, θα έπρεπε να βρούμε και άλλα μέτρα υποστήριξη τους. Κάτι ακόμα το οποίο ιδιαίτερα μας απασχολεί στην Ιρλανδία είναι το ζήτημα του πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει, χρησιμοποιήσει κανείς την έγωπροβατοτροφία ε, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Γιατί το λέω αυτό. Έχουμε μεγάλες περιοχές στην Ιρλανδία όπου προσπαθούμε να φυτέψουμε γρήγορα σοδιές οι οποίες πάρα πολύ σύντομα πρέπει να τις καταστρέψουμε και αυτό είναι ε, αρνητικό για το περιβάλλον. Ενώ ε, οι κτηνοτρόφοι που ασχολούνται με τα πρόβατα, που ασχολούνται με τη σταερήφια, έχουν αναγκαστικά μια πιο ε, βιώσιμη προσέγγιση στην κτηνοτροφία. Ε, επίσης, ε, οι άνθρωποι αυτοί βοηθάνε περιοχές στι οποίε διαφορετικά θα είχαν μαραζώσει οικονομικά. Ε, και κάτι ακόμα ιδιαίτερα για τη χώρα μου, υποστηρίζουν την Ιρλανδική γλώσσα. Σε αυτές τις περιοχές τι αγροτικές, τις κτηνοτροφικές, επιβιώνει η γλώσσα μας. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να τους βοηθήσουμε για το περιβάλλον, για την τοπική οικονομία, για τον τοπικό πολιτισμό, για τη γλώσσα την Ιρλανδική, ενώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθούμε να επιδιώξουμε εμπορικέ συμφωνίε με την ε, Αυστραλία, με τη Νέα Ζηλανδία, με χώρε με τι οποίε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ανταγωνιστούμε δεδομένων των τεράστιων εκτάσεων που έχουν. Ε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στο δικό τους επίπεδο. Επομένω, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, κονδύλια ευρωπαϊκά, ειδικά για τον τομέα αυτόν. Ευχαριστώ, Μισελ Νταντά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου προς την εισηγήτρια. Με κάλυψαν σε πολλά συνάδελφοι, δεν θα επαναλάβω λοιπόν κάποια σημεία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι υγειονομικό. Η εγωπροβατοτροφία και οι αντίστοιχες παραγωγές είναι ε, εκτατικές μορφές εκτροφής, όπου οι επαφές με την άγρια πανίδα είναι καθημερινές και άριθμες. Και ξέρουμε ότι η άγρια πανίδα σε μεγάλη κλίμακα κομίζει πολλές ε, ζωονόσους ή άλλες ασθένειες που θεωρούσαμε ότι είχαν εξελιχθεί. Βρουκέλωση, ε, φυματίωση. Πρόκειται για ε, νόσους που επηρεάζουν άμεσα την γεωργική παραγωγή και η προβατοτροφή ακριβώς πλήττεται από αυτή τη συνύπαρξη με την άγρια πανίδα. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε λοιπόν και αυτό το σκέλος. Και ίσως θα ήταν ενδιαφέρον και σκόπιμο η Επιτροπή μας, από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, να οργανώσουν μια δημόσια κρόση, ένα σεμινάριο για αυτό το θέμα. Δηλαδή, τις επαφές άγριας και η κόση της πανίδας ε, και τις ε, υγειονομικές συνέπειες αυτής της ε, επαφής. Κάποιος αναφέρθηκε και στην πανόλη των χείρων, ένα άλλο παράδειγμα τέτοιας επιζώτιας. Επίσης, ε, στην Γαλλία 10.000 ε, ε, ζώα έχουν χάσει, τη, έχουν χάσει τη ζωή τους από Γιατί λοιπόν να πάμε και εμείς στις Άλπεις στο σεμινάριο που θα γίνει για αυτό το θέμα. Ο Τζιμ Νίκολσον, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ράς Γκαρσία για την πολύ καλή της έκθεση. Όπως αναφέρθηκε, ε, η προβατοτροφία γίνεται κυρίως ε, στις πιο μειονεκτικές περιοχές, ε, λόφους, ορεινές περιοχές και μάλιστα σε περιοχές που καμία άλλη μορφή δραστηριότητας δεν θα ήταν δυνατή. Και ακριβώς λόγω της εκτεταμένης, εκτατικής τέτοιας κτηνοτροφίας με ελεύθερη βόσκηση έχουμε και σημαντική περιβαλλοντική αξία. Βέβαια, η εγωπαυροβατροφία είναι πολύ ευάλωτη στις δυνάμεις της αγοράς και συμμερίζουμε τις ανησυχίες των συναδέλφων, ε, ιδιαίτερα ε, τις ε, εκτενείς αγορές της Νέας Ζηλανδίας. Ε, φυσικά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις απέραντες ε, εκτάσεις βόσκησης της Νέας Ζηλανδίας με τα αντίστοιχα φωσκοτόπια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ε, της παραγωγής για μας. Ε, η αερινή αμνή είναι το προϊόν με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε αιχμή ευρωπαϊκής παραγωγής να μην επιτρέπουμε εκτεταμένες εισαγωγές από τρίτες χώρες. Και φυσικά ε, όποιος ήταν προβατοτρόφος και ξέρει ότι ε, ελάχιστα χρήματα ε, βγάζουν οι προβατοτρόφοι, γι' αυτό δεν έχουν επενδύσουν σε offshore σίγουρα. Και επίσης να λάβουμε υπόψη και τις συνέπειες του Brexit. Ε, θα, έχει συνέπειες στο Brexit όχι μόνο για όσους θα παραμείνουν, αλλά και για εμάς που αποχωρούμε γιατί ένα μεγάλο τμήμα των σφαγών γίνονται ε, πέραν των συνόρων του Ηνωμένου Βασίλειου. Οπότε το Brexit ε, και το θέμα του συνόρου θα επηρεάσουν πολύ και την απορροβατοτροφία. Επίσης, είναι σαφές ότι είχαμε μείωση 20% του αριθμού των ε, ποιμνίων και των, ζώων. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναχαιτήσει τέτοιου είδους πτώση, τέτοιου είδους μείωση. Τι, την παλιά εποχή είχαμε και για τις προβατίνες πρημοδοτήσεις και για τις ε, ε Τώρα έχουμε ε, ενισχύσεις ε, αναστραματική έκταση. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουν στις εκμεταλλεύσεις τους ε, ε αγελάδε ή προβατίνες για να λαμβάνουν το, ε, το πριμ τους. Προτιμούν να έχουν θυλάζουσες αγελάδε, που έχουν υψηλότερο, υψηλότερη πρημοδότηση. Οπότε αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα και στο μέλλον έχω σοβαρές ανησυχίες στην Σαβοία. Ε, ο κύριος Δαντά έχει πρόβλημα τους λύκους. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τους λύκους. Αλλά με τα, τον τρόπο που δίνονται χρηματοδοτήσεις. Ο κύριος Σεράου Σάντο. Σάντος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την ε, κυρία Ράνς Καρσία για την έκθεσή της και που πραγματικά μας κάνει εύκολη τη ζωή γιατί έκανε πολύ σημαντική προεργασία και ήδη βρισκόμαστε σε προηγμένο στάδιο της συζήτησης. Είναι σημαντική συμβολή της εγωπροβατοτροφίας στη διαφύλαξη της βιοπικιλότητας, όπως λέει και η κυρία Ρας Γκαρσία, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών ε, και της μετακίνησης ε, των ζώων ε, που εξεχυμάζουν σε άλλα Περιοχέ. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά, τα ειδικά χαρακτηριστικά των μεσογειακών βοσκοτόπων, όπως είναι το Μοντάδο στην Πορτογαλία, Ντέσσα, στην Ισπανία. Επίσης, θα πρέπει να διαφυλάξουμε την δραστηριότητα, δεδομένου ότι τέτοια κτηνοτροφία γίνεται σε απόμακρες μειονεκτικέ περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτε στην εγκατάλειψη, στην απερίμνωση και άλλο σημαντικό θέμα είναι η κατάρτιση των ποιμένων, που επισήμανε η κυρία Αγγιλέρα που είναι πραγματικά καταπληκτική ιδέα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια σταθερότητα των παραγωγών και της παραγωγής και καλό θα ήταν να απλουστεύσουμε το σύστημα ταυτοποίησης που είναι ιδιαίτερα επαχθές κυρίως για τους μικρής κλίμακος κτηνοτρόφους. Και να μην ξεχνούμε και τις επιθέσεις θηρευτών όπως λύκων ε, ή άλλων θηρευτών. Είναι ολέθριες οι συνέπειες στο ε, αριθμό των ερηφίων και των ε, αμνών. Θα πρέπει όχι μόνο να αποκαταστήσουμε τις ζημιές των κτηνοτρόφων, αλλά να επικεντρωθούμε και στην πρόληψη των επιθέσεων των θηρευτών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νέκοφ. Σας ευχαριστώ. <clears throat> Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με τον Έρικ οργανώσαμε συναντήσεις στη Νότια Γαλλία και στην Βουλγαρία οι οποίες έτυχαν θετικής υποδοχής. Κάτι που δεν αναφέρθηκε είναι ότι δεν υπάρχει ε, επαρκή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τις βέλτιστες πρακτικές. Κάτι ακόμα που διαπιστώσαμε από αυτές τις συναντήσεις είναι ότι χρειάζεται να, υπάρχουν σφαγεία κοντά στα βοσκοτόπια, κοντά στους κτηνοτρόφους. κτηνοτρόφοι δεν γνωρίζουν αναγκαστικά και ούτε μπορούμε να το αναμένουμε από αυτούς να γνωρίζουν πώς να προωθήσουν το προϊόν τους. Επομένω πρέπει να ε, υπάρχει κάποιος που θα τους βοηθήσει. Έχουμε τα συστήματα γεωγραφικής προέλευσης, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Χρειάζεται επίσης, κατά την άποψή μου, να, είμαστε πιο, να έχουμε μια προσέγγιση πιο ευέλικτη όσον αφορά τη στήριξη των ορεικνών περιοχών και ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που μας αναφέρουν οι παραγωγοί είναι ότι χρειάζονται ε, περισσότερους πόρους στις ορεινές περιοχές και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρέπει να το απαιτήσουμε εμείς αυτό. Και το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να φροντίσουμε το επίπεδο χρηματοδότησης που υπάρχει στη σημερινή κοινή πολιτική να διατηρηθεί ή ακόμα και να αυξηθεί. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σχάπ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και επίσης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την εκθεσή της. Ε, συνεργαστήκαμε στενά με την εισηγήτρια, με την ομάδα της και νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για ένα θέμα όπου νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στις βασικές αρχές. Όλοι συμφωνούμε ότι ο τομέας αυτός ε, κατά καιρού ε, χρειάζεται μία περαιτέρω όθηση για να αντιμετωπίζεται ως ένας τομέας όπου αναπτύσσονται σημαντικές δραστηριότητες. Ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω όσον αφορά την ε, υποστήριξη νομίζω ότι ήδη υπάρχουν ε, αρκετές μορφές ε, υποστήριξης ε, προς τους γεωργούς. 450 εκατομμύρια περίπου δαπανάμε κάθε χρόνο, κυρίως και ιδιαίτερα για να διασφαλίζουμε την παραγωγή στις περιοχές εκείνες όπου τα κράτη-μέλη θέλουν να διατηρήσουν την ε, εκτροφή εγών και προβάτων. Το δεύτερο που κάνουμε είναι πρόθεση στην εσωτερική αγορά αλλά και σε άλλες χώρες. Θα γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα εργασίας του 2018 ήδη προβλέπει σημαντική αύξηση των διατηθέμενων κονδυλίων για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να τονιστεί. Το τρίτο που είναι σημαντικό για εμάς είναι η αποκαλούμενη συνεργασία, ευρωπαϊκή συνεργασία καινοτομία. Υπάρχουν πολλές τεχνικές, ε, βέλτιστες πρακτικές. Μπορούμε να πούμε στους ε, γεωργούς πώς μπορούν να οργανώσουν καλύτερα την ε, εγώ προβατοεκτροφή. Ε, και για το μέλλον λοιπόν έχουμε στόχο τη βελτίωση όχι μόνο στον τομέα των προβάτων αλλά και για άλλους τομείς όπου νομίζω ότι καλύτερα μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τα προγράμματά μας ε, καινοτομίας. Σήμερα με την απόφαση που ελήφθη για τον κανονισμό Omnibus, νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τους γεωργούς να οργανωθούν καλύτερα. Ξέρετε ότι η θέση τους στην αλυσίδα αξιών είναι πολύ σημαντική. Το θέμα δεν είναι να έχουμε καλό και ποιοτικό κρέας, αλλά και πώς αυτό θα μπει στην αλυσίδα διατροφής πώς ε, θα πουλιέται καλό ποιοτικό κρέας ε, στα καταστήματα, θα φτάνει στους ε, καταναλωτές. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους παραγωγούς και για όλους που ακολουθούν μετά στην αλυσίδα μεταποίησης. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι και η διαφάνεια στην αγορά να έχουμε στοιχεία για την εξέλιξη της αγοράς, για την ανάλυση, αναλύσεις για τις ε, αγοράς. Εμείς αυτά τα προβάλλουμε. Meet, Go, Chip, Dash, ε, εκεί μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε και τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την αγορά. Σήμερα Είχαμε πολλές συζητήσεις ε, για τους ε, θηρευτές, ε, για το θέμα των λύκων. Πράγματι, αυτό απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς και όλα αυτά τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για αποζημίωση. Τα κράτη-μέλη έχουν στη διάθεσή τους πολλά τέτοια μέτρα και είμαι σίγουρος ότι τα μέτρα αυτά θα χρησιμοποιηθούν κατά το μέγιστο. Κατά τα άλλα, επιτρέψτε μου να εκφράσω και μία προειδοποίηση. Ξέρετε, πρέπει να εργαζόμεθα μέσα στο εφιστάμενο πλαίσιο. Η οδηγία προβλέπει κάποια ευελιξία όσον αφορά στη διαχείριση των ζημιών ε, θα ήθελα λοιπόν όλοι μας να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο αυτή την ευελιξία ε, και αυτό από κοινού και με άλλες ομάδες, παραδείγματος χάρη ε, με αυτή για το περιβάλλον. Γιατί χρειαζόμαστε συνένεση για όλα αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα δεν είναι μόνο γεωργικά, δεν παίζει ρόλο μόνο γεωργία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και την υποστήριξη του ευρύτερου κοινού για οτιδήποτε κάνουμε. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή τη την έκθεση. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας. Ο τομέας ε, είναι πολύ ελκυστικός. Ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα θέματα. Ας συνεχίσουμε λοιπόν και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Σχάπ για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, το λόγο έχει η κυρία Ράνς. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας βοηθά και με την οποία συνεργαζόμαστε για το θέμα αυτό. Καταρχήν, είναι εκτενής ο κατάλογος των θεμάτων για τα οποία συμφωνούμε γενικώς. Το τελευταίο ζήτημα που έθιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο οποίο όλοι συμφωνούμε είναι το θέμα των θηρευτών. Ήμασταν πολύ γενναιόδοροι απέναντι στου θηρευτέ ε, από περιβαλλοντική άποψη, υπερβολικά γενναιόδοροι στα θεσμικά όργανα. Έτσι όμω βλάπτουμε του παραγωγικού μα τομεί με την υπερβολική γενναιοδορία που δείξαμε για του θηρευτέ. Ε, στην οδηγία για τα ενδιατήματα ή στο ψήφισμα που μα ανέφερε η κυρία Αγγιλέρα, δεν δείξαμε τη δέουσα κατανόηση προς τον παραγωγικό μας κλάδο. Οι επιθέσεις από αρπακτικά και θηρευτές αυξάνονται συστηματικά. Ξεκινήσαμε να είναι περιθωριακές και τώρα δημιουργούν σοβαρές πια ανησυχίες λόγω της συχνότητάς τους. Δεν πρέπει μόνο να προσπαθούμε να αποκαθιστούμε τις ζημιές. Χρειαζόμαστε και προστατευτικά και προληπτικά μέτρα γιατί φαίνεται ότι ιδιαιτεράχθηκε μέχρι στιγμή η ισορροπία μεταξύ θηρευτή και παραγωγή. Αν θέλουμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ του περιβάλλοντος και της εκτινοτροφικής παραγωγής, θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο ελαστικοί. Επίσης, ε, χαρμόσυνη ήταν η είδηση της ε, έγκριση του όμνιμπους και του διαχωρισμού του γεωργικού σκέλους. Βέβαια, κάποια σημεία θα τροποποιηθούν στην ψηφοφορία του όμνιμπους στην Ολομέλεια, Πάντως ευτυχώς ε, το γεωργικό σκέλος ε, έχει εγκριθεί και ε, φυσικά με τις τροπολογίες θα αλλάξει κάπως. Περιμένω και τις τροπολογίες και για τη δική μου έκθεση. Το θέμα των διεθνών εμπορικών συμφωνιών μας επηρεάζει. Η Νέα Ζηλανδία είναι μείζων παραγωγός, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη θέση της το Brexit, η αποχώρηση του μεγαλύτερου παραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίση να ληφθεί υπόψη και να λάβουμε υπόψη και, ότι, το έλλειμμα που έχουμε. Δεν είμαστε αυτάρκεις, αλλά θα πρέπει να προσπίσουμε το, τον παραγωγικό μας ιστό και να ενισχύσουμε την παραγωγή και τον κλάδο. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το σημαντικό περιβαλλοντικό ρόλο και την περιβαλλοντική αξία αυτής της εκτροφής. Ε, είναι ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά αυτή τη εκτροφή. Είναι αναντικατάστατη εγώ προβατοτροφία. Το είπε και η κυρία Σέρρα. Το θέμα του, της εκαθάρισης των δασών από τα βοσκοτόπια χάθηκε με το Natura 2000 ε, γιατί δεν μπορούν πια οι ιδιοκτήτες των δασών να κάνουν δασοκομική χρήση όπως μπορούσαν στο παρελθόν. Και μάλιστα αυτή η προβατοτροφία καθαρίζει το δάσος, οπότε είναι και πολύ χρήσιμη και φιλοπεριβαλλοντική και έχει και μία ε, φάση, ε, μία διάσταση πρόληψης ε, των δασών ή δασοπροστασίας. Επίσης, θα πρέπει να γίνει κάποια διάκριση, γιατί μερικές φορές η προβατοτροφία μπορεί να είναι εντατική, αλλά κατά κανόνα ο κλάδος είναι εκτατικής εκτροφής, μάλιστα σε μειονεκτούσες, μειονεκτικές περιοχές, απόμακρες, ορεινές, με πολύ χαμηλό επίπεδο. Και έτσι αναγκάζονται ο πληθυσμό να παραμείνει σε αυτές τις αγροτικές περιοχές με μεγάλες αντικσότητες και πολύ δυσκολότερους ε, δυσκολότερες βιωτικές συνθήκε από τις πόλεις και παρόλα αυτά οι άνθρωποι παραμένουν εφόσον έχουν κίνητρα για να ασχοληθούν με την εγωπροβατοτροφία. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση στην εκτατική εκτροφή ιδιαίτερα σε ε, αγροτικές περιοχές στην Ήπεθρο. Ε, επειδή η έκθεση πρωτοβουλία έχει κάποιους ε, περιορισμούς ως προς την έκτασή της, γι' αυτό δεν μπορούσα να είμαι υπερβολικά εξαντλητική. Ε, το θέμα των γυναικών, του ρόλου των γυναικών σε αυτή την εκτροφή, το τονίσατε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και το δίκτυο γυναικών κτηνοτρόφων που με βοήθησε στη σύνταξη της έκθεσης που πραγματικά έχουν ικανότητες και έχουν δικτυωθεί και όλα. Ελπίζω να μας ακούν, θα ήθελα να τους απευθύνω χαιρετισμό και να αναγνωρίσουμε φυσικά το ρόλο των γυναικών και σε αυτό το είδος εκτροφής. Ευχαριστώ τον κύριο Ντόρφμα και πολύ σωστά μιλήσατε για το μπημένα και τα χαρακτηριστικά της ειδικής αυτής εκτροφής. Οπότε να μην χάνουμε την εικόνα του βοσκού και τις σημαντικές ε, δεξιότητες που θα πρέπει να έχει. Μερικές φορές ε, οι νέοι κτηνοτρόφοι ε, βρίσκονται σε πλήρη άγνοια όταν ξεκινούν την παραγωγή και χρειάστηκε να εκμεταλλευτούν την πλούσια πείρα και τις γνώσεις των πιο παλέμαχων εκτροφέων. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε το σημαντικό ρόλο των ποιημένων και περιμένω τη σχετική τροπολογία σας για την κατάρτισή τους. Σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, επίσης συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις πρακτικές και να βελτιώσουμε και την παρουσίαση, την τελική παρουσίαση του προϊόντος στον καταναλωτή, ώστε να γίνει ελκυστικό αυτό το κρέας και για νέους καταναλωτές η κατανάλωση μειώνεται γιατί ε, δεν είναι πια δεκτικός ο καταναλωτής. Παλιά αγοράζαμε το αρνί ολόκληρο. Ε, τώρα είναι αδιανόητο να αγοράσει κάποιος ε, έστω και μισό αρνί και να χρειάζεται να τρώει το ίδιο κρέας μέρες ολόκληρες. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έφαση και στις νεοειδικοποίησεις για να προσελκύσουμε περισσότερους καταναλωτές. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους. Θα συνεχίσουμε τη, τις εργασίες μας. Ξεκινά η διορία για την υποβολή τροπολογιών και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το φιλικό και θερμό εγκάρδιο κλίμα μεταξύ μας για να έχουμε αγαστή συνεργασία, κάτι που είναι προς όφελος του κλάδου, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αυτό το κλάδο για να παραμείνει η ύπεθρος με κόσμο, με αγρότες. Σα ευχαριστώ να χαιρετήσω και εγώ το δίκτυο γυναικών κτηνοτρόφων, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντική η συμβολή του και μάλιστα η παρουσία των γυναικών στο, στην κτηνοτροφία είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο και χαίρομαι που μέσω, των, ε, μέσω κοινωνικής δικτύωσης μεταφέρουν τι ανησυχίε τους. 27 Νοεμβρίου Μία το μεσημέρι λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και τον Ιανουάριο έχει προβλεφθεί η έγκριση της έκθεσης αυτής. Περνάμε στο σημείο 7, την μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκθεση πρωτοβουλίας ε, είναι και αυτή ε, που έχουν ε, αναλάβει για την γνωμοδότηση οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, ο κύριος Καπούτο, που όμως απουσιάζει, θα τον αντικαταστήσει όμως ο κύριος Αντριέ, που θα μας παρουσιάσει τον προβληματισμό αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας ο Ερίκ Αντριέ. Ευχαριστώ Κλάρα. Αντικαθιστώ εδώ τον Νικολά Καπούτο που προτείνει άρδιν μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων και νέους μάλιστα ίδιους πόρους για να μειωθεί ε, το, ε, η συνεισφορά από το ΑΕ που ήταν 67,5 το 2016 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, είναι προφανές ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων ε, δεν λειτουργεί και περιλαμβάνει περίπλοκους ε, και διαφανείς μηχανισμούς διορθωτικούς. Και μάλιστα κάθε χρόνο έχουμε ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών. Τα συμπεράσματα τη ομάδα υψηλού επίπεδου για του ίδιου πόρου με πρόεδρο τον Μάριο Μόντι περιλαμβάνει νέε προτάσει που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, όπω για παράδειγμα μία μεταρρύθμιση του ίδιου πόρου του ΦΠΑ ή ένα, μεταρρύθμιση στο φόρο του συστήματο εμπορία εκπομπών ή φόρο στο διοξίδιο του άνθρακα, στι μεταφορέ, στην ηλεκτρική ενέργεια και στα έσοδα τη ενιαία ψηφιακή αγορά. Ο Νικολά λοιπόν καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να αντιλήσουν τα κατάλληλα συμπεράσματα από την έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους και να, να εξετάσουν την σκοπιμότητα και το πόσο είναι εφικτό τέτοιες συστάσεις να εφαρμοστούν για να κάνουν πιο αυτόνομη, προβλέψιμη και πιο ε, δίκαιη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων είναι απαραίτητη για να χρηματοδοτηθούν πρόσφατε προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετανάστευση, ασφάλεια, ε, και ε, να αντισταθμίσουμε και την απώλεια 12 δισεκατομμυρίων ε, λόγω του Brexit. Επίσης, θα πρέπει να αντισταθμίσουμε την μείωση πόρων που προτείνει ο κύριος Έτιγκερ για, στο έγγραφο προβληματισμού για τα μελλοντικά οικονομικά της Ένωσης, γιατί με τέτοια συρρήκνωση του κοινωτικού προπολογισμού θα επηρεάσει σημαντικά και την γεωργική πολιτική. Και μάλιστα είναι σημαντικό και οι γεωρικοί δασμοί να διασφαλιστούν στο μέλλον, όπως προτείνει η ομάδα υψηλού επίπεδου για τους ίδιους σπόρους, γιατί και αυτοί οι γεωρικοί δεσμοί είναι σημαντικός απλός ε, ίδιος Τη ε, της Ένωσης. Θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Επίση, να μην ξεχνούμε την προστιθέμενη αξία τη ΚΑΠ ε, στην ενίσχυση τη επιστηστικής ασφάλεια, τη μακροπρόθεσμη επιστηστικής ασφάλεια. και να επιμείνουμε στην ανάγκη διασφάλιση των γεωργικών δικαιωμάτων στα δημοσιονομικά και στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τους και ηγητές. Πρώτα το λόγο έχει ο κύριος Κούσμιουκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση του κυρίου Καπούτου είναι καλή και μας αρέσει. Καλό θα ήταν όμως στην γνωμοδότησή μας να τονίσουμε πιο έντονα τη σημασία που έχει η κοινή γεωργική πολιτική για την επιστημιστική ασφάλεια αφενός και αφετέρου για τη σταθερότητα των ε, τιμών των τροφίμων. Γιατί αυτό το θέμα ε, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες, όπως ε, ε, η γαλακτοκομική παραγωγή στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία επηρεάζουν ε, πολύ την, ε, τις τιμές του βουτύρου και κυρίως την αύξηση του τιμού του βουτύρου που είναι απαράδεκτη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Επίσης, το πρόβλημα με την αύξηση των τιμών των αυγών λόγω του φιπρονίλ και της καταστροφής σημαντικού αριθμού των πτηνών, των ε, οτόκων ορνήθων, κάτι που οδήγησε σε ε, αύξηση της τιμής των αυγών. Και αυτό είναι ε, ακατανόητο και απαράδεκτο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Να τονίσουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η ΚΑΠ για την εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών των τροφίμων, που είναι βασικό χαρακτηριστικό της ΚΑΠ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέτορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι είναι ε, ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα ο προϋπολογισμός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε σχέση με τους ίδιους πόρους. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα πρόσδεκτο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναλαμβάνονται οι ευθύνε για να υπάρχει σωστή διαχείριση ε, και στα έσοδα και στα έξοδα. Πάντως πρέπει να ε, προετοιμαστούμε για τις μελλοντικές προκλήσεις διότι τα κράτη-μέλη ε, δεν, έχουν, δεν αντιμετωπίζουν όλα τις ίδιες οικονομικές εξελίξεις. Αν υπήρχε ένας δείκτης ΦΠΑ, θα ήταν δύσκολο για ορισμένα κράτη να μεταφέρουν, τις, να μετακυλούν τη συνεισφορά τους ή να εμβάζουν τη συμφορά τους στον κοινωτικό προεπλογισμό. Αν δούμε το ΑΕΠ ε, υπάρχουν τεράστιες ε, διαφορές ε, από 60.000 μέχρι 120.000 Υπάρχουν ε, πολλές ε, διαφορές ε, και στις τιμές. Όσον αφορά λοιπόν τη γεωργία και το σύστημα των πληρωμών, οι πληρωμές διαφέρουν μέχρι και 70%. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το θέμα των ιδίων πόρων είναι πολύ σημαντικό και οφείλουμε και εμείς να το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά. Η πρόταση που έχει κατατεθεί να υπάρχει ένα συντελεστής. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ επιφυλακτικά, γιατί οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντενανό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι έχει βάλει το δάκτυλο επί τύπο τον ήλωνο συνάδελφος Νικολά. Είναι ναι, ε, το ζήτημα των ιδίων πόρων αιώνιο θέμα που το συζητούμε από τότε που δημιουργήθηκε η νέα αγορά. Κάθε τόσο το συζητούμε και μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει μια λύση. Πιστεύω ότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βρει μια λύση. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να, έχουμε, να εγκρίνουμε τον προπολογισμό των εξόδων χωρίς να έχουμε μια αντίστοιχη άποψη για τα έσοδα. Ίσως το Brexit να είναι να μπορεί να φέρει κάτι καλό ε, πέρα από το, τα άσχημες επιπτώσεις του και αυτό το καλό να είναι η αναθεώρηση του συστήματος των ιδίων πόρων. Πράγματι έχουμε νέες πολιτικές ε, στον τομέα της ε, καταπολέμησης της ενεργείας, της μετανάστευσης, της άμυνας που πρέπει να τις χρηματοδοτήσουμε αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις παραδοσιακές πολιτικές, ε, τις, τα διαρθρωτικά ταμεία, την κοινή γεωργική πολιτική, τις ε, πολιτικές συνοχής που ε, φροντίζουν και ενισχύουν την ίδια την δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως δεν θα πρέπει να τις παραμελήσουμε ή να της, ε, να παραμεληθεί η δημόσια χρηματοδότηση αυτών προς όφελος ε, της ιδιωτικής. Χρειάζεται λοιπόν να τις ενισχύσουμε αυτές τις πολιτικές οι οποίες ε, επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν πρέπει να τις εγκαταλείψουμε. Αντιθέτως, η κοινή γεωργική πολιτική και αυτές οι πολιτικές συνοχή είναι αυτές τις οποίες πρέπει να ενισχύσουμε. Ευχαριστώ κύριο Σουλάναγκα. Στο πρώτο σημείο, στην αρχή ακριβώς της έκθεσης, ζητείται μια εκφάθρον αναθεώρηση του συστήματος των ιδίων πόρων και να βρεθούν και νέε νέες πηγές ιδίων πόρων. Ναι, αυτό ακούγεται καλό, αλλά στην πραγματικότητα θα δώσει ακόμα μεγαλύτερε εξουσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα πολύ απλό τρόπο να καλύψουμε το κενό που δημιουργεί το Brexit και αυτό είναι να αυξηθεί η συνεισφορά που βασίζεται στο ακαθαριστό εγχώριο προϊόν, εάν αυτό το θέλουμε. Όμω αυτό που θα ε, ήταν το αποτέλεσμα αντί να προσπαθεί κανείς να βάλει περισσότερο νερό σε ένα βαρέλι που έχει διαρροή, θα ήταν καλύτερα να φροντίσει να, να ε, επιδιορθώσει τη διαρροή. Και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές διαρροές. Έχουμε ε, περιπτώσεις ε, παραγωγών ή ανθρώπων οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την κοινή γεωργική πολιτική ενώ δεν θα έπρεπε. Αντί λοιπόν να ρίχνουμε νερό σε αυτό το δοχείο που στάζει, θα πρέπει να κλείσουμε τις τρύπες του ένα πρόβλημα που έχουμε στην Ιρλανδία είναι ότι το καθόριστο ε, εισόδημα ε, ε, υπολογίζεται με τρόπο μη αξιόπιστο. Λέγεται ότι η Ιρλανδία έχει ξεπεράσει την οικονομική κρίση. Πώς τα κατάφερε αυτό. Όταν και, και, και, και, Έχουμε αναφέρει μάλιστα μια αύξηση του ΑΕΠ 28%. Αυτό στην πραγματικότητα ε, ε, είναι πλασματικό. Ε, δεν υπήρξε καμία τέτοια μεγέθυνση του ΑΕΠ, δεν υπήρξε τέτοια ανάκαμψη της Ιρλανδικής οικονομίας. Πώς θα το, υπολογίζει κανείς αυτό. Δεν θα πρέπει να βρούμε μια, ένα σύστημα υπολογισμού του, του εισοδήματο, το οποίο να είναι πολύ καλύτερο και πολύ πιο αποτελεσματικό από το υπολογισμό του ΑΕΠ δεδομένων των συνοπιών που έχει αυτός, αυτή, αυτός ο υπολογισμός. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, θα συμφωνήσω με τον κύριο Φλάναγκαν ε, να υπάρξει άλλη μία παράγραφος γιατί αυτή τη στιγμή οι διπόροι προκύπτουν μόνο από, τους δασμούς, από επιβολή, από το ΦΠΑ ε, και από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Τώρα, αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους ζητάει να υπάρχει μία νέα φορολογία και τώρα πλέον οι γεωργοί θα φορολογούνται για τα εγωπρόβατά τους μια νέα μορφή φορολογίας. Το ίδιο ισχύει και για τους ε, καλλιεργητές οποροκυπευτικών. Αυτοί ε, χρηματοδοτούνται για τις καλλιέργειές τους ε, και μετά όμως θα πρέπει να φορολογούνται. Αυτά πρόκειται να έρθουν στο μέλλον. Ελπίζω λοιπόν να τα χαρείτε πάρα πολύ, να ευχαριστηθείτε. Κύριε Άγνιο, εσείς πάντως δεν πρόκειται να το απολαύσετε, γιατί είστε Βρετανός, οπότε από τη στιγμή που θα αποχωρήσετε, ελάχιστα θα απολαύσετε καθόλου το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ ένα ειρωνικό σχόλιο όπως εσείς. Έχουμε ολοκληρώσει με τους συναδέλφους. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα των ιδιών πόρων. Σημειώνουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι αναφερθήκατε στην ομάδα υψηλού επίπεδου ε, με πρόεδρο τον κύριο Μόντι που υπέβαλε πολύ ενδιαφέρουσε προτάσεις για τους μελλοντικούς ιδίου πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γνωρίζετε ότι όχι μόνο για τους λόγους που αναφέρθηκαν, αλλά και λόγω του Brexit ε, και την αποχώρηση ενός σημαντικού καθαρού συνεισφορέα ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις χώρες που ήταν ε, προτεργάτης του, του μηχανισμού των εκτόσεων και με την κατάργηση αυτού του μηχανισμού και των σταδιακών εκτόσεων θα χρειαστεί μεταρρύθμιση. Όχι γιατί θα χάσουμε μεγάλο αριθμό κονδυλίων, αλλά και γιατί η διάρθρωση του παλιού συστήματος χρήζει μεταρρύθμισης. Δεν έχουμε ακόμη αποκρισταλώσει τις ιδέες μας. Το Μάιο του 2018, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της. Πάντως, ακούσαμε πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις και από τον εισηγητή για νέους ίδιους πόρους που θα εξεταστούν στην εσωτερική συζήτηση που θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, Αναφερθήκατε πολύ στον παράγοντα του ΑΕ, του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος. Πρόκειται για ένα σύστημα που εισήχθη για να εξορροπηθεί το σύστημα μεταξύ των κρατών μελών και το ΑΕ ε, τη χάνει ιδιαίτερη υποστήριξη στα κράτη-μέλη, γιατί θεωρούν ότι έτσι γίνεται ε, δίκαιη κατανομή του μεριδίου του στον κοινοτικό προπολογισμό, λαμβάνοντα ω ε, γνώμονα το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ε, βέβαια, στις συζητήσεις ε, για το νέο σύστημα ιδίων πόρων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οποιοδήποτε νέο σύστημα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για δίκαιο επιμερισμό του φόρτου ή του, του, του άχθους στο κοινοτικό προϋπολογισμό των κρατών μελών και να μην είναι ανισότιμα τα μερίδια τους. Μια και ο κύριος Καπούτα απουσιάζει σήμερα, ο Ερίκ Αντριέ θα ολοκληρώσει αυτή τη συζήτηση εκ μέρους του εισηγητού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που υπέβαλα για την έκθεση και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεταρρύθμιση των ίδιων πόρων ε, ε, θα πρέπει να γίνει και μάλιστα κατεπηγόντως και εκβάθρων, γιατί 9 με 13 δισεκατομμύρια θα είναι το κενό το χρηματοδοτικό από το Brexit. Αλλά έχουμε και νέες προκλήσεις που επίσης ε, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την ίδια βάση το 1% της εθνικής συνεισφοράς στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αν δεν αλλάξουμε τον, κανόνα το 1% και αν δεν επιταχύνουμε τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων, πιστεύω όπως και ο εισηγητής ε, και όχι περικόπτοντας φυσικά την ε, πολιτική συνοχή στην κυνηγιορική πολιτική. Χωρίς εκβάθρο μεταρρύθμιση δεν πρόκειται να επιλύσουμε το πρόβλημα. Τώρα πια έχουμε στριμωχθεί. Έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και δεν μπορούμε με τεχνάσματα να μετακυλούμε στον επόμενο χρόνο την ε, τήρηση των υποχρεώσεων μας. Θα πρέπει επιτέλους να μεταρρυθμίσουμε και τον κανόνα των 1% και τη χρηματοδότηση των νέων προκλήσεων με άρδεν μεταρρυθμίση των ιδιών πόρων. Η έκκληση του Νικολά Καπούτο και η παραπομπή στι συστάσει τη ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου δείχνουν ότι θα πρέπει από κοινού να επιταχύνουμε οπωσδήποτε τι συζητήσει για τη μεταρρύθμιση του στήματο των ιδιών πόρων. Μάλιστα, ολοκληρώθηκε η συζήτηση η προθεσμία για τι τροπολογίε για την γνωμοδότηση αυτή λήγει στι 27 Νοεμβρίου, μία το μεσημέρι, όπως και ε, η προθεσμία για την προηγούμενη έκθεση. Και περνάμε στο επόμενο θέμα και θα αλλάξει και πάλι ο Πρόεδρος στη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και πάλι πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας, εμείς έχουμε τη γνωμοδότηση, πρόκειται για ένα θέμα αλληλένδετο με το προηγούμενο και είναι σημαντικό που τα συζητούμε εκ παραλλήλου. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας που είναι η κυρία Σοφία Ριμπέιρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ε, σας μεταφέρω τη μεγάλη αβεβαιότητα που νιώθουν ε, οι γεωργοί μας ε, και αυτό είναι το κύριο θέμα της γρομοδότησης μου. Ε, ζητούν ε, αύξηση του γεωργικού προϋπολογισμού, αύξηση την, της, ε, των άμεσων ενισχύσεων χωρίς χρηματοδότηση, ε, επιπλέον ποσά για τη διαχείριση των κρίσεων και καταπολέμηση των αθέμετων εμπορικών πρακτικών. Θεωρώ ο, θεμελιώδη ανάγκη να ενισχύσουμε τα συστήματα στήριξης και της γεωργίας και των νέων γεωργών και κυρίως των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των μειονεκτικών περιοχών της Ένωσης, διαφυλάσσοντας το πρόγραμμα ΟΣΕΙ και τη χρηματοδότησή του. Ε, βέβαια, μέχρι στιγμής έχει φτάσει στα όρια του ΟΣΕΙ και ο πενιχρός προπολογισμό του. όλα αυτά φυσικά είναι στα χέρια μας, στα χέρια σας, αλλά θα πρέπει να δείξουμε πυγμή εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας, προσπίζοντας την Ευρωπαϊκή Γεωργία, την ιστορία της και προσπίζοντας και τους Ευρωπαίους Γεωργούς, γιατί ο γεωργικός μας κλάδος υφίσταται από τις σημαντικότερες επιθέσεις ε, της ιστορίας μας. Η κοινή γεωργική πολιτική, που είναι η πιο παλιά πολιτική της Ένωσης, είχε θεμελιώδη ρόλο στην επιστημιστική ε, αυτάρκεια και ασφάλεια του της Υπήρου μας μετά το τέλος του πολέμου. Επίσης, ε, ε, σίγουρα έχουν αλλάξει οι καιροί, αλλά οι γεωργοί τώρα χρειάζονται τη γεωργή, την βοήθειά μας, γιατί το γεωργικό του εισόδημα έχει μειωθεί τόσο πολύ και έχει γίνει τόσο αβέβαιο, που πραγματικά δεν ξέρουν τι αύριο τους περιμένει. Ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και τις αθέμετες εμπορικές πρακτικές. Θα τι άλλες κρίσεις χρειαζόμαστε για να έχουμε μια στέρεη νομοθεσία. Οι, κυρίως ε, οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές μας ε, βρίσκονται στο έλεος τους γιατί ε, δεν στηρίζουμε την γεωργική τους οικονομία και τις κοντινές αλυσίδες ανεφοδιασμού με αποτέλεσμα να έχουμε εγκατάλειψη της υπαίθρου και απερίμωση αυτών των περιοχών που ήδη ήταν φτωχές. Και ε, μερικές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς να εξετάζουμε τον αντίκτυπό τους για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές με εμπορικές ε, συμφωνίες που προκαλούν προβλήματα χωρίς να προβλέπουν επαρκείς αντισταθμίσεις. Όταν ε, κερδίζουμε θα πρέπει όλοι να κερδίζουμε και όχι να κερδίζουμε μερικής βάρος κάποιων άλλων. Έχουμε το γεωρικό προϋπολογισμό στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας τριακονταετίας ε, ακόμη και με τις περιβαλλοντικές αιρεσιμότητες. Και τώρα θέλουν να προσθεθούν και νέες αιρεσιμότητες. Και μάλιστα με το Brexit είναι μάλλον ζωφερές οι προοπτικές. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ ότι οι ενισχύσει τη ΚΑΠ είναι απαραίτητε για να έχουμε ποιοτικά γεωργικά προϊόντα σε προσιτέ τιμέ. Επίσης δεν θα πρέπει να φοβόμαστε στην προάσπιση του γεωργικού προϋπολογισμού. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε από κοινού με τους και να καταλήξουμε σε μια άρτια στη βαρύ έκθεση, ε, επανεπιβεβαιώνοντας και διατρανώνοντας την αποφασιστικότητά μας να προασπίσουμε τους Ευρωπαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους και προσβλέπω στη συνεργασία σας για να το καταφέρουμε. Ευχαριστώ Σοφία. Η Κλάρα Αγγιλέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ως και ηγήτρια της ομάδας μου για την γνωμοδότηση αυτή, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, τη Σοφία, γιατί πραγματικά η γνωμοδότησή της στα ένα καλό σημείο αφετήριας. Με ανησυχούν κάπως ε, τα, τα θέματα των προθεσμιών γιατί είναι σημαντικό να ολοκληρώσουμε τη γνωμοδότησή μας πριν την ε, έγκριση της ε, αρμόδιας κατουσίαν επιτροπής, της έκθεσης της Επιτροπής Προϋπολογισμών δηλαδή. Με προβληματίζει λοιπόν ε, το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Γιατί όταν μιλούμε για προπολογισμό έχουμε πολλά διακυβεύματα και στην Επιτροπή Γεωργίας. Γιατί μπορούμε να χαράζουμε πολιτικές, αλλά αν δεν τις τροφοδοτούμε με το, τα απαραίτητα κονδύλια και χρηματοδοτικούς πόρους, θα είναι ε, μία τρύπα με στο νερό. Θέλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε μία ισχυρή κοινή πολιτική, Φυσικά κάποιες πτυχές της θα πρέπει να αλλάξουν και να μεταρρυθμιστούν, αυτό είναι αναφυσβήτητο, αλλά θα πρέπει, αμή τι άλλο, ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ να παραμείνει άθικτος. Κάτι άλλο που με προβληματίζει και προέκυψε και στη συζήτηση με τον Επίτροπο Έτιγκερ είναι η προβλέψιμη επανεισαγωγή της χρηματοδότησης. Επίσης, στην γνωμοδότησή μας θα πρέπει να αντιταχθούμε στην πιθανότητα συγχρηματοδότησης στον πρώτο πυλώνα, στις ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε μια κοινή γεωργική πολιτική, ο πρώτος πυλώνας θα πρέπει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν θεσπίσουμε τη συγχρηματοδότηση και στον πρώτο πυλώνα, τότε επανερχόμαστε σε κρατικές πολιτικές που θα διαμορφώνουν τους στόχους μας. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε τον πρώτο πυλώνα αποκλειστική ε, κοινοτική αρμοδιότητα με αποκλειστική κοινοτική χρηματοδότηση χωρίς ε, δυνατότητα συγχρηματοδότηση. Μόνο έτσι θα έχουμε διαφοροποιημένη ε, κοινή γεωργική πολιτική που δεν θα υπακούει σε κρατικούς σχεδιασμούς. Επίσης, πέραν των αρχών της ΚΑΠ και σε άλλες περιόδους, η κοινή γεωργική πολιτική έκανε τέτοιε προσπάθειε, συνέβαλε τόσο πολύ στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, στην προστασία του περιβάλλοντο, που δεν μπορούμε να την αγνοούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι ο προπολογισμό στηρίζει μόνο μία οικονομική ε, γεωργική δραστηριότητα, αλλά συμβάλλει και στην περιβαλλοντική αξία και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της γεωργίας και άλλα προστατεύει και το κλίμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το εξάρουμε. Επίσης, το σημείο 6 μιλάτε για την ανάγκη χρηματοδοτικού και νομικού πλαισίου. Αυτό ε, θα πρέπει να γίνει στη δική μας κοινοβουλευτική θητεία και ελπίζω, όπως υποσχέθηκε ο Επίτροπος Χόγκαν, το Μάιο να υποβάλει το χρηματοδοτικό και νομικό πλαίσιο για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ώστε να καταπολεμήσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Δεν είναι κακό που το αναφέρουμε, γιατί η πολιτική δεσμεύση του Επιτρόπου Χόγκαν δεν νομίζω ότι αρκεί. Δεν ξέρω αν είναι σημαντικό να έχουμε πολλά μέτρα. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι τα μέτρα να είναι δίκαια και σαφή και να εξηγούν την ανάγκη που έχουμε στον 21ο αιώνα να συνεχίζουμε τις επιδοτήσεις. Και φυσικά είναι σημαντικό ε, να τύχει της υποστήριξης μας αυτή η γνωμοδότηση. Έχουμε ένα νέο δασμό που επιβλήθηκε στις επιτραπέζιες ε, ισπανικές ελιές αυτό τον έδωσμο τον επέβαλαν οι Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί θεωρούν ότι οι γεωργικές ενισχύσεις της ΚΑΠ προκαλούν dumping στις Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό ε, πρόσθεσαν νέο εμπορικό δασμό για τις ισπανικές επιτραπέζιες ελιές 6%. Αυτή είναι μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στην κοινή γεωργική πολιτική και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι από κοινού να την προστατεύσουμε όπως της αξίζει. Ο κύριος Κούσμιουκ, σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γνωμοδότησης για την περίπλοκη αυτή σύνθετη γνωμοδότηση που υπέβαλε για την μελλοντική χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής και να προσθέσω και ένα επιπλέον επιχείρημα ε, υπέρ της προάσπισης ε, και της διατήρησης αμή άλλο του ισχύοντος επίπεδου χρηματοδότησης. Όπως είπε και η κυρία Αγγιλέρα, έχουμε νέες υποχρεώσεις ε, που αναλαμβάνουν οι Γεωργοί με την κοινή γεωργική πολιτική. Την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της φύσης, του φυσικού τοπίου. Όλα αυτά συνιστούν νέες υποχρεώσεις για τους γεωργούς ε, που κατοχυρώνονται από την κοινή πολιτική και φυσικά θα πρέπει να προβλέψουμε κατάλληλη χρηματοδότηση για να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις. Στο σημείο 4 η εισηγήτρια ε, μιλά για τις άθικτες άμεσες ενισχύσεις ε, και για να αποφευθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ε, να μην προβλεφθεί η χρηματοδότηση. Εγώ θα ήθελα να πω ως Πολωνός ότι αυτό το, αυτή η διαδικασία της εναρμόνισης των επιδοτήσεων μεταξύ παλιών και νέων χωρών ε, και το σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα θα πρέπει να εξαλειφθεί γιατί δημιουργεί άδικη μεταχείριση μεταξύ των παλιών και νέων χωρών. Και φυσικά στις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ε, το κόστος παραγωγής και μεταποίησης ήταν χαμηλότερο. Αλλά στο μεταξύ έχουμε ε, πλησιάσει στα επίπεδα των υπολείπων χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Και μάλιστα για την προστασία των φυτών, ε, το κόστος φυτοπροστατευτικών προϊόντων τώρα είναι χαμηλότερο στη Δυτική Ευρώπη από ό,τι στην Κεντρική και Ανατολική. Οπότε αυτή η διαφοροποίηση που υπήρχε δεν δικαιολογείται πια. Ε, και μάλιστα όλα τα γεωργικά προϊόντα κυκλοφορούν στην ίδια αγορά γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε θετικές ε, και ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού. Αυτή η εξομοίωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές και σχετική κατάθεση, ε, τροπολογία θα καταθέσω και εγώ. Ο κύριος Ντενανό. Σας ευχαριστώ. Χρειάζεται σταθερότητα και ενίσχυση η ευρωπαϊκή αγροτική οικονομία. Και χρειάζεται μια στήριξη η οποία να είναι διαρκής. Και η χρηματοδότηση από την ΚΑΠ θα πρέπει να είναι υψηλή. Έχουμε ανταγωνιστές, μεγάλα κράτη, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα και η Συγήτρια έχει δίκιο να υπογραμμίζει την υποκρισία των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα αυτό. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε πολλαπλές κρίσεις ε, υγειονομικές, την κλιματική αλλαγή, οι οποίες ε, διακινδυνεύουν τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά αναφέρει η κυρία Ριμπέρο στην εκθεσή της, θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε, θα πρέπει να φροντίσουμε να ενισχυθεί η ΚΑΠ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. συμφωνούμε όλοι ότι το Brexit ε, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα ε, και στον τομέα της κοινή γεωργικής πολιτικής και υπάρχουν δύο δυνατότητες είτε να μειώσουμε γενικότερα τον προϋπολογισμό και να πείσουμε τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν τα ίδια το κενό που θα προκύψει στο μέλλον, αλλά βέβαια το γεγονός ότι τώρα η κοινή γεωργική πολιτική παίρνει το 38% των πόρων ε, σε σχέση με το 60% που έπαιρνε πριν από κάποια χρόνια, ίσως ε, τώρα να έχει βρεθεί μια λύση και να μπορεί η κοινή γεωργική πολιτική να αντιμετωπίσει μόνη της τα προβλήματα γιατί υπάρχουν κρίσεις σε, σε πάρα πολλούς άλλους τομείς και ίσως τα κράτη-μέλη μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στο να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις σε άλλους τομείς ε, πολιτική γειτονία ε, ή ε, να, αντί να δίνουν χρήματα στην κοινή γεωργική πολιτική. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο και σκέπτομαι Πότε ε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των εισαγωγών. Έχω κατά νου θέματα και περιθώρια, παραδείγματο χάρη μέγιστη υποστήριξη ε, σε μία και μόνο εκμετάλλευση ίσως θα πρέπει να βάλουμε όρια από 100 μέχρι 150 χιλιάδες αναεκμετάλλευση οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις ε, μπορούν να διαφοροποιηθούν, ε, μπορούν να αναπτύξουν εναλλακτικέ δραστηριότητε. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και κάτι άλλο. Ε, άδικο σύστημα πληρωμών. Αν επιτρέψουμε στους λιανέμπορους και στους χοντρέμπορους να ορίζουν τις τιμές που οι ίδιοι επιθυμούν, τότε δεν θα συμβάλλουμε στο να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες στις αγροτικές περιοχές. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Ο συνάδελφός μου από την Πολωνία ανέφερε ότι έχει έρθει, έχει, έχει φτάσει πια η στιγμή έτσι ώστε να καταργηθούν οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα παλιά και τα καινούργια κράτη-μέλη. Μία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας είναι ο κώδικας ε, των νομικών πράξεων και όσον αφορά στα γεωργικά και τα περιβαλλοντικά μέτρα θα πρέπει να έχουμε μία ενιαία στάση. Βέβαια οι πληρωμές διαφέρουν και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Νομίζω ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου έτσι ώστε να αρχίσουμε να προβάλλουμε διαφορετική προσέγγιση. Κατά την άποψή μου η διαχείριση των κρίσεων είναι σημαντική. Ε, πολλά κράτη δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση και αυτό το στοιχείο θα πρέπει να είναι σημαντικό στις ε, πολιτικές μας. Εξάλλου, οφείλουμε και στους ε, δημόσιους διαγωνισμούς και εκεί να επιβάλλουμε ειδικές φορές. Κάρτη, Σα um, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινή γεωργική πολιτική αυτές οι διαφορές ενισχύονται και νομίζω ότι έχει έρθει πια η στιγμή για μας ε, για να αναγνωρίσουμε, να δεχτούμε ε, τα πραγματικά ωφέλη της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, δηλαδή που ωφελείται η Ευρωπαϊκή Ένωση από όλα αυτά τα ωφέλη. Εγώ πιστεύω μεγάλο όφελος είναι ότι διασφαλίζουμε ποιοτική, ποιοτικά τρόφιμα και ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχει ανάπτυξη της υπέτρου των περιφερειών και μπορούμε να είμαστε και σίγουροι ότι τα καλύτερα τρόφιμα του κόσμου έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε λοιπόν πώς θα επιμερίζει το προπλογισμό για να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι οφείλουμε τα κονδύλια να τα κατευθύνουμε ε, σε μικρομεσαίους ε, γεωργούς γιατί πραγματικά υπάρχει τεράστιες, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στο πώς επιμερίζονται τα κονδύλια. Και νομίζω ότι Πρώτα απ' όλα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αυτή η Επιτροπή αλλά και άλλοι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι οφείλουμε να αλλάξουμε την όλη δυναμική μέσα στην κοινή γεωρική πολιτική. Και κάτι άλλο. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να προστατευτεί ο προϋπολογισμός της κοινή γεωρική πολιτικής. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν περίπου 4 ε, δις ευρώ ε, που θα λείψουν Εάν λοιπόν θέλουμε να πουλήσουμε συσταγωγικά στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό με την επιβολή φόρων ή επιβάλλοντα τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τι εισφορέ του. Δεν νομίζω ότι αυτό θα τύχει ευρεία υποστήριξη. Εγώ θέλω να σα πω, οφείλουμε να προστατεύσουμε την κοινή γεωργική πολιτική και ε, σε άλλου τομείς, δαπάνες ε, για την ασφάλεια, ε, για στρατιωτικού εξοπλισμού, εκεί μπορούν να υπάρξουν περικοπέ. Αυτό πρέπει εμεί ω Επιτροπή να προβάλλουμε και αυτό θα τύχει ευρεία αναγνώριση. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρο, Τώρα έχουν μιλήσει σκιώδης. Τώρα η υπόλοιπη είναι Ο κύριος Σάντος. Ευχαριστώ Παόλο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Σοφία Ριμπέιρο για την γνωμοδότησή της που έχει στρατηγική σημασία για το μέλλον και τη διαβεβαιώ ότι θα τη βοηθήσω και θα τη στηρίξω όσο μπορώ. Χρειαζόμαστε κάποια σαφήνεια στη Γεωργία γιατί αν συγκρίνουμε με άλλες οικονομικές δραστηριότητες βλέπουμε ότι διατρέχει σημαντικό κίνδυνο και λόγω κλίματος, λόγω επιζωτιών, λόγω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά. Αυτό επίσης ε, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα των γεωργικών τιμών ουσιαστικά αφήνει ε, ξεκρέμαστο το γεωργό ή μπορεί να τον αφήσει ξεκρέμαστο από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς να εξασφαλίζει καν το προστοζήν. Γι' αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε τον, ε, γεωργικό, τον αγροτικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί συμβάλλει πολύ και στην επιστηστική ασφάλεια και στη διαφύλαξη της χωροταξίας και του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή γεωργική πολιτική επαρκώς ε, πρικοδοτημένη ώστε να δίνει μια μελλοντική προοπτική για τους αγρότες και κίνητρα για να παραμείνουν στη δραστηριότητά τους. Οπότε το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποδείξουμε και να δείξουμε πυγμή και αποφασιστικότητα στην προάσπιση του γεωρικού μας προϋπολογισμού. Επίσης θα πρέπει στο μέλλον να ενισχύσουμε την θετική διαφοροποίηση των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, των μειονεκτικών περιοχών. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα να σα υπενθυμίσω στι αρχέ του έτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έκρινε θετικά το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙ, που είναι σημαντικό πρόγραμμα για τις εξόχως απόκεντες περιοχές, Μαδέρα και Αζόρες, και έκρινε ε, πολύ θετική την αποτελεσματικότητα και τη σημασία του για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική συνοχή. Τέτοιου είδους μηχανισμοί είναι ε, περίτρανη απόδειξη της ε, θετικής συνέπειας που έχουν τα κοινοτικά κονδύλια και μάλιστα κινητοποιήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να αναδείξουμε τη σημασία αυτού του εγγράφου, να προσπίσουμε το, τη διατήρηση του προγράμματος ΠΟΣΕΙ και να ενισχύσουμε μάλιστα την πρικοδότησή του για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Ευχαριστώ κύριο Σκαλινόφσκι. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας να την ευχαριστήσω γιατί τόνισε την ανάγκη όχι μόνο διατήρησης του ισχύοντος ορίου της ΚΑΠ αλλά και την ενίσχυσή του εν ώψη των κυκλικών κρίσεων των νέων προκλήσεων, την ανάγκη σημαντικών εργαλείων για να καταπολεμήσουμε αυτή την αβεβαιότητα και τη φοβερή αστάθεια των τιμών. Βέβαια, μιλάτε ότι λέτε ότι περίπου 4 δισεκατομμύρια το έτος θα είναι το χρηματοδοτικό κενό του Brexit, για να μην μιλήσουμε για τις νέες προκλήσεις ε, που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν, όπως είναι η ασφάλεια, το μεταναστευτικό, η μεταναστευτική κρίση και εκεί έχουμε, θα έχουμε ρίκνωση του προπολογισμού κατά άλλα δισεκατομμύρια που ίσως επηρεάσουν ε, και τον γεωργικό προϋπολογισμό. Ε, Επίσης, ε, θα θέλαμε να γίνει δεκτή η ε, διατήρηση της ε, εθνικής συνεισφοράς για να μην συρρυκνωθεί ο προπολογισμό, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη να αυξήσουν την συνεισφορά τους στον κοινοτικό προπολογισμό για να διαφυλάξουμε και την ΚΑΠ μεταξύ άλλων. Ε, επίσης, λέτε ότι θα πρέπει να η σύγχρηματοδότηση για τις άμεσες ενισχύσεις και μάλιστα όχι σε προαιρετική βάση γιατί δεν θα γίνει δεκτό. Θα πρέπει να δώσουμε τα κράτη-μέλη να, να αναπληρώσουν τις ε, ζημίες που θα προκληθούν από το Brexit στη χρηματοδότηση της ΚΑΠ ε, αλλά ε, στο επίπεδο των περικοπών μόνο. Κάτι τέτοιο δεν θα πειράσει τον ανταγωνισμό και οι γεωργίδες σκέφτονται από πού προέρχονται τα χρήματα. Τους ενδιαφέρει πραγματικά να γίνεται αποκατάσταση των ζημιών και να ε, λαμβάνουν τις πληρωμές που δικαιούνται. Οπότε, σας παρακαλώ ε, να υπάρχει δυνατότητα εκτάκτως συγχρηματοδότησης, όχι, ε, όχι σε προαιρετική βάση, αλλά ώστε να μην αυξηθούν οι ζημιές στην χρηματοδότηση της ΚΑΠ μόνο για αυτή την αντιστάθμιση. Α, επικίνδυνο λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Αντρία και μετά η κυρία Ερά. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Σοφία Ριμπέιρου για την έκθεση και τι προτάσει της. την υψηλή ποιότητα, Εγώ δεν θα ήθελα να δούμε η κοινή αγροτική πολιτική να είναι τελικά μια παράπλευρη απώλεια της υποχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ε, επιδιώξεών της. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να μπορεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Και αυτό είναι πραγματικά που θα ε, εξαρτηθεί, που διακυβεύεται μάλλον στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι ως Ήπειρος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχουμε τους απαιτούμενους πόρους και δεν, βρίσκουμε, δεν βρούμε τους μηχανισμούς για να έχουμε τους απαιτούμενους πόρους. Δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ούτε τις σημερινές ούτε τις νέες, τις μελλοντικές προκλήσεις εάν δεν ε, ενισχύσουμε ε, τις πολιτικές που βρίσκονται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η καινή γεωργική πολιτική και οι πολιτικές συνοχής. γεωργία δεν είναι ένας τομέας της οικονομίας ίδιος με τους υπόλοιπους. Ε, πρόκειται για την πηγή για των τροφίμων μας, πρόκειται για το περιβάλλον, πρόκειται για τη δημόσια υγεία. Και επομένως χρειάζεται μια πραγματικά ε, ουσιαστική δημόσια πολιτική ε, στήριξη της γεωργίας. Βεβαίω δεν μπορούμε να στηρίξουμε κάθε έναν παραγωγό ξεχωριστά, αλλά χρειάζονται μέτρα, αντίστοιχα με τα σημερινά, μέτρα κανονιστικού χαρακτήρα που να φροντίζουν την υγεία των καταναλωτών, αλλά επίσης και μέτρα για την ε, ενίσχυση της ε, συγκεκριμένων περιοχών που μπορεί να μειονεκτούν. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την προσπάθεια να έχουμε πιο, πιο κοντά στο πολίτη, την, την, την ε, μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών, με το να χάσουμε τον ευρωπαϊκό μας προσανατολισμό. Επομένως, για αυτόν τον λόγο είμαι εναντίον της συγχρηματοδότησης. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι πιο μακρόπνο, όχι απλώς τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά τα επόμενα δέκα χρόνια, να σκεφτούμε πώς θέλουμε να εξελιχθεί η γεωργία μας. Λαμβάνοντα υπόψη ότι το πληθυσμό του πλανήτη θα αυξηθεί στα νέα δισεκατομμύρια, θα πρέπει να βρούμε πώς θα ε, ε, τραφεί. Είναι ζήτημα λοιπόν διατροφικής ασφάλειας και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα τα απαραίτητα για να την ε, εξασφαλίσουμε αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία ράνς Γκαρσία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τη Σοφία Ριμπέρο για το έργο της και να υπενθυμίσω ότι ζητά από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις εθνικές τους συνεισφορές στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το σύστημα αυτό είναι και το πιο δίκαιο. Έχω την αίσθηση ότι οι χώρες που έχουν περισσότερα έσοδα θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο και χώρε που έχουν λιγότερα λιγότερα. Και αυτό είναι πιο διαφανές. Ε, γιατί με τους φόρους ε, ε, θα διαμαρτυρηθούν οι πολίτες ότι τους κοστίζει πιο πολύ από ό,τι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βγούμε όλοι χαμένοι. Με την αύξηση των εθνικών συνεισφορών θα έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια από ότι με την αύξηση των φόρων. Αν όλοι θέλουμε μια ισχυρή κοινή πολιτική με εξασφάλιση του του προϋπολογισμού τους. Πριν από λίγο μιλήσαμε για τα εγωπρόβατα. Ε, θέλουμε ταυτόχρονα ισχυρή πεθρό, ισχυρή γεωργία και κτηνοτροφία, προστασία του περιβάλλοντος, ποιοτικά τρόφιμα σε προσιτές τιμές. Αν θέλουμε όλους αυτούς τους στόχους θα πρέπει να αυξήσουμε ε, τις εθνικές συνεισφορές στον κοινοτικό προπολογισμό για να κρατήσουμε άθεκτο τον γεωργικό προϋπολογισμό γιατί αναμένονται περικοπές ε, στο γεωργικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει όμως να εξορθολογήσουμε την ΚΑΠ, γιατί αν τα κράτη-μέλη συμβάλλουν ε, και στις πληρωμές του, του, πρώτου πυλώνα, θα αρχίσουν να συμμετέχουν και αποφάσεις. Οπότε δεν θα αποφασίζουμε εμείς, αλλά τα κράτη-μέλη θα αποφασίζουν για τη μορφή της ε, κοινή γεωργική πολιτικής και θα την επανεθνικοποιήσουμε έτσι. Άρα θα χάσουμε τις κοινοτικέ αρμοδιότητες. Θέλουμε μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική ε, η ΚΑΠ θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι από τι πιο ισχυρέ πολιτικές ε, του κοινοτικού προπολογισμού, γιατί είναι από τις πολιτικές που πιο κοντά βρίσκονται στον Ευρωπαίο πολίτη. Η κυρία Μίλλερ, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η επαρκής χρηματοδότηση είναι και η πραγματική βάση για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να συμφωνήσουμε από αυτού ότι στο μέλλον θα ενταθούν κατά πολλοί απαιτήσει όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τον έλεγχο τη ασφάλειας παραγωγής τροφίμων, παραδείγματος χάρη στον τομέα των ε, ζυζανιοκτώνων. Ε, εδώ οι γεωργοί θα αντιμετωπίσουν όλο και περισσότερα προβλήματα, ε, θέματα τα οποία πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την κοινή γεωργική πολιτική. Οι γεωργοί χρειάζονται την ασφάλεια και γι' αυτό με αυτή την έκθεση πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Πέρα από την απλούστευση, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τη χρηματοδότηση. Ε, το ύψος του προπολογισμού θέλουμε να το διατηρήσουμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια κυρίως για το σημείο υπαριθμών 2 το οποίο προσέθεσε, δηλαδή μέσα στην Ευρώπη να υπάρξουν εκστρατείε ενημέρωσης για το τι μπορεί να επιτευχθεί με όλα αυτά τα χρήματα. Διότι η ΜΚΟ και η προστασία, όσοι ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, δεν επιθυμούν να δοθούν αυτά τα κονδύλια. Θεωρώ ότι ο σωστός δρόμος είναι να υπάρξει μια εκστρατεία ενημέρωσης. Και κατά τα άλλα επιθυμώ οι άμεσες πληρωμές να διατηρηθούν και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να επεκταθεί σε 7 χρόνια. Εκ μέρου ε, του σκιώδη συγητού μας, ε, του κυρίου Τάκουλο, που οποίος δυστυχώς έχει ε, ασθενήσει, εμείς θα στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον θα καταθέσουμε προτάσεις που θα ενισχύσουν τη γεωργία και θα εκπέμψουν και ένα χειρό μήνυμα προς την κοινή γνώμη. Ο κύριος Μισελ Νταντάν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεσή της. Ας μην ξεχνούμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική έχει ως πρώτο στόχο να εξασφαλίζει την διατροφική μας ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Και γνωρίζουμε ότι αυτό δεν επιτυγχάνεται, δεν μπορεί να επιτυχθεί μάλλον, παρά μόνο εάν υπάρχει η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία καταφέρνουν να παράγουν περισσότερα ε, οποροκυπευτικά φρούτα, άλλα τα οποία καταφέρνουν καλύτερα στα σιτηρά. Επομένω αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών έχει επιτρέψει τελικά στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να απολαμβάνει τη μεγαλύτερη διατροφική ασφάλεια από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη. Ωστόσο, πρέπει να βρούμε και τρόπους να ε, έχουν ένα ικανοποιητικό εξόδημα όλοι οι γεωργοί. Εάν διαιρέσουμε το σύνολο των γεωργικών ενισχύσεων με τον αριθμό των ε, γεωργικών μονάδων και το δούμε και πόσο φτάνει αυτό ανά μήνα, ε, δεν είναι ικανοποιητικό το γεωργικό εισόδημα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν. Το 95% των προϊόντων έρχεται από το 20% των μονάδων του γεωργικών, είναι οι πιο παραγωγικές και είναι αυτές οι οποίες εξάγουν επίσης. Μίλησε πριν ο συνάδελφος για το, την, την, ότι ο πληθυσμό του πλανήτη θα φτάσει στα 9 δισεκατομμύρια και πρέπει να βρούμε πώ θα διατρέφεται. Ε, δεν πιστεύω ότι αυτό αναλογεί στην Ευρώπη. Πρέπει να βρούμε πρώτα απ' όλα τρόπου για να εξασφαλίσουμε τη διατροφική ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, και ε, ξεχνούμε ότι ε, η κοινή γεωργική πολιτική είναι απαραίτητη σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, ιδιαίτερα τη Μεσόγειο. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε οποιοδήποτε προσπάθεια η οποία πάει να μας διχάσει και οποιαδήποτε προσπάθεια επανεθνικοποίησης αυτών των πολιτικών με όποιον τρόπο και αν αυτή διατυπώνεται, είτε διατυπώνεται ας πούμε με την ε, υιοθέτηση εθνικών, πολιτικών, εθνικών κριτηρίων, γιατί αυτό θα ε, μας κάνει να οπισθοχωρήσουμε και στην πραγματικότητα θα επηρεάσει ε, δυσμενώς τους πλέον ευαίσθητους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ κύριο Φλάνεγκαν. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή. Συμφωνώ με αυτά που λέξαν στο σημείο 5. Πρέπει όμως να προτείνω μία αλλαγή. Δηλαδή εκεί λέει ότι ε, να υπάρξει άμεση υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη. Και πιο κάτω γίνεται λόγο στο φάκελο. Ε, νομίζω πρέπει να πούμε ότι υπήρξε ε, κάποια βοήθεια για όσους χρειάζονται, βρίσκονται σε ανάγκη. Άρα δηλαδή πρέπει να πούμε να συνεχιστεί η βοήθεια. Είναι πιο σωστό το να συνεχιστεί. Το 4% των άμεσων πληρωμών ε, μοιράζεται σε πάνω από μισούς. Ε, ε 250 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η βοήθεια. Σύμφωνα με το σημείο 2 θα πρέπει να υπάρξει ε, εκστρατεία ενημέρωσης. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα αν είχαμε σωστή κατανομή. Αλλά αυτή τη στιγμή η εκστρατεία ενημέρωσης είναι ότι έχουμε ανθρώπους όπως ο Λάρι Γκότμαν και την βασίλισσα της Αγγλίας που παίρνει ε, βοήθεια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τι είδους εκστρατεία έχετε κατά νου. Να βελτιώσουμε τη ζωή των πλουσίων και να γίνουν οι φτωχοί πιο φτωχοί. Δεν μπορεί να υπάρξει εκστρατεία όταν η κατάσταση είναι αυτή που περιέγραψα. Εγώ δεν έχω δουλέψει σε γεωργική εκμετάλλευση. Είμαι άνθρωπος της πόλης, αλλά βλέπω όλα αυτά τα ωφέλη που προέρχονται από την κοινή γεωργική πολιτική. Ο πατέρας μου ήταν ξυλουργός ε, όταν δούλευε και ε, είχε άμεση σχέση με τους γεωργούς. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τα χρήματα της γεωργίας είναι πολύ χρήσιμα. Κυρίως αν δει κανείς το Brexit και τις επιπτώσεις για τις συνοριακές περιοχές ε, χωρίς ε, να δοθούν τα χρήματα στους γεωργούς βλέπουμε ότι με το να υπάρχει ένα σύστημα όπου θα μειωθούν οι πληρωμές θα βιώσουμε καταστάσεις όπου οι εκατομμυριούχοι θα πάρουν και άλλα εκατομμύρια. Αλλά οι χώρες που θα πληγούν από το Brexit αυτές δεν θα λάβουν τίποτα. Ως ετούτου η κοινή γεωρική πολιτική ε, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλή αλλά αυτή τη στιγμή ε, δεν κατανοώ πώς είναι δυνατόν να πληρώνουμε εμείς για τα διαμάντια της Βασίλισσας. Απαράδεκτα πράγματα. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι οι προκλήσεις είναι τεράστιες και εν ώψη του Brexit και εν ώψη των νέων δημοσιονομικών υποχρεώσεων. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση για να εξασφαλίσουμε τα επαρκή κονδύλια για την κοινή γεωργική μας πολιτική. Επίσης, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την αποδοχή της γεωργίας στα μάτια της κοινή γνώμης. Ε, η γεωργία είναι μειονότητα στο συνολικό πληθυσμό. Είναι πολύ μικρό ποσοστό, γι' αυτό και ο κόσμος ε, ε, δεν καταλαβαίνει τη θέση των γεωργών. Γίνεται πολύ κακή διαφήμιση των γεωργών, ιδιαίτερα όταν μιλούμε πολλά για φυτο, πολύ για φυτοφάρμακα και λοιπάσματα. Και είναι δύσκολο να προσυτεριστούμε το κοινό υπέρ της ε, γεωργίας και γεωργικής πολιτικής. Μας μην ξεχνούμε όμως ότι χάρη στους γεωργούς εξασφαλίζουμε την επιστηστική μας ασφάλεια. Η γεωργία μας είναι σημαντική και για την υγεία μας και για το περιβάλλον μας. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε τον προϋπολογισμό. Θέλουμε ενδελεχή και ανοιχτή συζήτηση. Να μην ξεχνούμε και την καινοτομία στη γεωργία και την κτηνοτροφία και να βοηθήσουμε και τους νέους γεωργούς, να τους δώσουμε κίνητρα για να ασχοληθούν με τη γεωργική δραστηριότητα και να εξασφαλίσουμε και υψηλή παραγωγικότητα ώστε να έχουν υψηλά εισοδήματα. Θα πρέπει και οι νέοι γεωργοί να βρουν στη γεωργία μία προσοδοφόρο δραστηριότητα, αλλιώς ε, δεν θα έχει νόημα να ασχοληθούν με αυτήν. Ε, έχουμε πολλές ε, προκαταρκτικές δράσεις ε, για τα ΕΦΗ χωριά στη Σλοβενία, πολύ Τώρα έχουμε επιχειρηματικά μοντέλα στις πόλεις, αλλά γιατί να μην εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο και στα χωριά. Η ανάπτυξη πέθρου είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές και να αδράξουμε και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα της υγείας και αλλού. υπάρχουν δυνατότητες ε, για την ανάπτυξη πέθρου, τονίζοντας το ρόλο της στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Επίσης, ε, να δώσουμε κίνητρα στους γεωργούς, ε, ώστε να ασχοληθούν όλο και περισσότερο με μια προσοδοφόρο γεωργική δραστηριότητα, για να τους αρκούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Α, ο κύριος Χόισλινγκ μάλλον έχει το ίδιο επίθετο με τον συνάδελφο, γι' αυτό έδωσε το λόγο κατά λάθος στον κύριο Χόισλινγκ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα να πω και εγώ μερικά λόγια. Πρώτα απ' όλα, αρκετοί από εσάς ε, καταθέσατε προτάσεις ε, για το πώς θα εξελιχθεί η πολιτική αυτή στο μέλλον. Εγώ θα σας παραπέμψω στην επόμενη Τετάρτη, όταν ο Επίτροπος κύριος Χόγκαν εδώ σε αυτή την Επιτροπή ε, θα παρουσιάσει την ε, ανακοίνωση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και είμαι σίγουρος ότι εκεί θα υπάρξει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Όσον αφορά τώρα τα θέματα που σχετίζονται με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και με τον γεωργικό προϋπολογισμό. Αρκετοί από εσάς ε, αναφέρατε τη λέξη αβεβαιότητα, το γεγονός ότι ο τομέας ε, χρειάζεται σταθερότητα. Συμφωνεί απόλυτα από αυτού η Επιτροπή. Ε, βέβαια γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις. Θα υπάρξει περικοπή διότι ένας σημαντικός καθαρός συνεισφορέας εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν πολιτικές άλλες που χρειάζονται μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Ο κύριος Οτιγκέρο ο Επίτροπος, το έχει πει αυτό επανειλημμένο, ότι αυτά τα δύο από κοινών τα συνδυάσει αποτελούν πολύ μεγάλη πίεση για το μέλλον του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και προφανώς και οποιασδήποτε άλλη, οποιασδήποτε πολιτικής δαπανών. Αρκετοί από εσάς ε, θίξε το θέμα της συγχρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην ανακοίνωσή της ε, του Ιουνίου σχετικά με το μέλλον της χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Επιτροπή προβάλλει μια σειρά θεμάτων για το πώς τα κενά ε, που μεταξύ έχουν προκύψει, πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν και πώς θα χρηματοδοτηθεί και η ΚΑΠ μετά το Brexit. Η ε, συγχρηματοδότηση είναι ένα θέμα που υποβλήθηκε για συζήτηση, τίποτα άλλο όμως δεν έγινε, η Κομισιόν δεν τοποθετήθηκε, σίγουρα όχι ο Επίτροπος κ. Χόγκαν. Πάντως υπάρχει η όλη συζήτηση γιατί με τον τρόπο αυτό ε, θα τεθεί το θέμα πώς ε, θα αντιμετωπιστούν ενδεχόμενε περικοπές στην κοινή και γεωργική πολιτική και οι επιπτώσεις τους ε, στους ε, νέους γεωργούς. Αναφερθήκατε και στον αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν πρόκειται για χρήματα, για τον προπολογισμό, αλλά για τις σωστές, σωστές συνθήκες έτσι ώστε η γεωργία να μπορεί να ανταγωνίζεται τους άλλους τομείς στην αλυσίδα με μεγαλύτερη δικαιοσύνη θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να βοηθήσει κανείς τον γεωργικό τομέα έτσι ώστε αυτός να βρεθεί σε ισχυρότερη θέση. Πιστεύω ότι η εξωτερική σύγκληση που αναφέρατε πολλοί από εσάς που ε, καταρχήν είναι η διαφορά ανάμεσα στις πληρωμές, στις ενισχύσεις, καταβολή πληρωμ... ενισχύσεων που υπάρχει. Ε, είναι διαφορετικές αυτές οι ενισχύσεις στα διάφορα κράτη-μέλη και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το θέμα δεν είναι ανάμεσα στην Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη και οι διαφορές αυτές δεν έχουν απαραίτητα σχέση μόνο με τα παλαιότερα αποκαλούμενα νέα κράτη-μέλη. Ε, κάποιος ε, αναφέρθηκε στο ότι η, τα κονδύλια για την ΚΑΠ από 60% πήγαν στο 40%. Πράγματι, στη δεκαετία του 70 η ΚΑΠ είχε πολύ μεγάλο ποσοστό στον προπολογισμό. Τότε βέβαια ο προπολογισμό ήταν πολύ πιο μικρός και λιγότερες πολιτικές. Τότε ας πούμε δεν υπήρχε πολιτική συνοχή. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει κανείς τώρα ότι ο προπολογισμό της ΚΑΠ μειώθηκε ουσιαστικά στη διάρκεια των ετών. Ε, θα πρέπει περισσότερο να πούμε ο προϋπολογισμός παρέμεινε ο ίδιος σταθερός ε, βεβαίως ε, ε, προφανώς επειδή άλλαξαν οι συσχετισμοί άλλαξε και το ποσοστό της ΚΑΠ κατά τα άλλα εγώ δεν λέω, δεν τοποθετούμε επί του ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Ξέρετε όμως ότι τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν επ' αυτού. Και ε, θα υπάρξουν δύσκολες συζητήσεις ε, για το μέλλον του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τη διάρκεια, το χρονικό διάστημα, ε, άκουσα με ενδιαφέρον ότι πολλοί τάσσονται και υπέρ της αυξημένης ε, χρονικής διάρκειας για το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό πρέπει να μπει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η θέση του Κοινοβουλίου έτσι είχαμε καταλάβει επιθυμεί να είναι μικρότερο το χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο ε, νομίζω ότι επ' αυτού θα υπάρξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα σαφέ ότι επιθυμούμε να υπάρχει σταθερότητα στι δαπάνε, κυρίω για την ΚΑΠΑ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τέλο, μερικοί από εσά αναφερθήκατε στι ε, περικοπέ, ε, στα κατόφλια, ε, ανώτατα κατώτατα όρια για τις πληρωμές υπάρχει ένα σχετικό έγγραφο για το πώς μπορούν να κατευθύνονται πιο στοχευμένα οι επιδοτήσεις. Και ανακεφαλαιώνοντας θέλω να πω ότι τελικά ε, θα υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση όχι μόνο για την ΚΑΠ αλλά έχοντας ε, κατά νου και τον ευρύτερα, το ευρύτερα δύσκολο πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη πίεση θα ασκηθεί, ε, πρέπει να το γνωρίζουμε, να είμαστε ρεαλιστές και νομίζω περισσότερο από ποτέ έχει έρθει η στιγμή να έχουμε μια πολιτική ε, που να μπορεί κανείς να τη στηρίξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε την Επιτροπή και τώρα το λόγο έχει η Σοφία Ριμπέρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους τις παρατηρήσεις που έκαναν. Και χαίρομαι γιατί σε γενικές δραμές, συνολικά, φαίνεται να συμφωνούν με τις κυριότερες προτάσεις που έχω υποβάλει. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ΚΑΠ δεδομένων των πολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων που έχουμε σήμερα. Πράγματι, θα υπάρξει πίεση για περικοπές στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, οι ανάγκες των ε, γεωργών ε, αυξάνονται και οι υποχρεώσεις τους στην ποιότητα ε, των προϊόντων τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν προσπαθούμε να θρέψουμε όλο τον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ε, μειωθεί η ΚΑΠ ή να περάσουμε όλα τα προβλήματα στους παραγωγούς. Δεν μπορούμε από τη μια να αυξάνουμε τις ε, απαιτήσει και από την άλλη να μην έχουμε πόρους για να μπορούμε να τις υλοποιήσουμε. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα του επίπεδου των τιμών. Και επίσης ε, έτσι θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη σύγκληση και εδαφική και κοινωνική συνοχή όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών που είναι σημαντικό να υπάρχει τέτοια συνοχή αλλά και ε, στο εσωτερικό ε, του κράτους μέλους μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της ίδιας χώρας. Οπότε θα πρέπει να έχουμε διαφοροποιημένη μεταχείριση εκεί που όντως υπάρχουν διαφορές και ιδιαιτερότητες. Και θα ήθελα να επισημάνω κάποιες νέες ε, προκλήσεις όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές που θα πρέπει να μετριάσουμε δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος με τις νέες απαιτήσει που θέτουμε να αυξάνουμε τη γραφειοκρατία για τους γεωργούς. Θα πρέπει και εδώ να επιδιώξουμε την απαραίτητη ισορροπία. Επίσης, ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις εμπορικές συμφωνίες ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τρόπο όμως που θα προστατεύει τη γεωργία ώστε να μην γίνει η Γεωργία ο φτωχό συγγενή αυτών των διεθνών συμφωνιών εμπορικών συναλλαγών. Θα πρέπει να τη δώσουμε το βάρο που της αξίζει και σε οικονομικό επίπεδο στο παγκόσμιο προσκήνιο. χωρί να αμελούμε και να ε, ξεχνούμε τη σημαντική κοινωνική διάσταση που έχει επίση η Γεωργία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των απολογιών είναι 27 ε, Νοεμβρίου, 3 η ώρα. Και ε, στις 23 Ιανουαρίου ε, θα ψηφίσουμε για την έγκριση της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ όλους και σε 5 λεπτά οι συντονιστές.